Okay. Yeah, yeah. Do la parola. Do la parola al vicepresidente. Δίνω το λόγο στον Αντιπρόεδρο Βαζεβόφσκι. Κύριε, κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, η Πολωνία έχει πληγεί από μια τρομερή τραγωδία και σίγουρα θα έχετε ακούσει για, την, για το τραγικό αυτό αεροπορικό δυστύχημα του Σαββάτου κατά τη διάρκεια του οποίου ο πρόεδρος της Πολωνίας, η πρώτη κυρία της Πολωνίας σκοτώθηκαν. Επίσης, ο πρώην πρόεδρος μας σε εξορία στο Λονδίνο, στο παρελθόν, και πάνω από 90 υψηλοί αξιωματούχοι, υπουργοί, μέλη του Γενικού Επιτελείου. Έχασαν και αυτή τη ζωή τους. Οι ιερείς, λοιπόν, στρατιωτικοί και μέλη της οικογένειας των ατόμων αυτών που είχαν χάσει πριν από 70 χρόνια στο Κατίν του οικείους τους έχασαν τη ζωή τους. Ταξίδευε το αεροπλάνο αυτό προς το Κατίν, όπου πάνω από 22.000 Πολωνοί αξιωματικοί εξοντώθηκαν από τις μυστικές υπηρεσίες της Σοβιετικής Ένωσης μετά από εντολή του Στάλιν. Και οι, εκεί οι οικογένειες ε, κάποιες από τις οικογένειες αυτών των ατόμων έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την αεροπορική καταστροφή. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή για την Πολωνία και είμαστε όλοι συγκλονισμένοι μετά από αυτό το γεγονός. Εάν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να σας ζητήσω να κρατήσουμε τώρα ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της τεράστιες αυτής αεροπορικής καταστροφής σε μνημή του Πρόεδρου της Πολωνίας και όλων των ατόμων που το συνόδευαν. Grazie Vicepresidente Vacevoschi, grazie a tutti voi. Questa tragedia ci ha colpito tutti. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο, κύριο Βασεγόφσκι. Αυτή η τραγωδία έπληξε όλους μας. Εγώ ήμουνα την προηγούμενη στη Βαρσοβία, όπου συνάντησα τον ε, Υπουργό Βαζαβίνσκι. Πρόκειται για μια τεράστια τραγωδία για όλους. Ξεκινάμε τη συνεδρία της Επιτροπής μας. Καταρχήν έγκριση της ημερήσιας διάταξης, αν δεν έχετε τίποτα, εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Όπως ανακοίνωσα και την προηγούμενη εβδομάδα, πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε την κυρία Ελίζαμπεθ Γέγγελ, η οποία θα μας αναφέρει τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται ως πειραματόζωα και η συνέχεια που θα δοθεί. Μετά θα εξετάσουμε το τμήμα το σχετικό με τον προπολογισμό για την ΚΑΠ και μετά παρουσία του Ντάσιαν Σιόλος θα συζητήσουμε την έκθεση του George Lyon σχετικά με το μέλλον της κάποια το μετά το 2010. Αν δεν έχουμε τίποτα άλλο, έχουμε, να σας πω ότι έχουμε διερμηνία προς όλες τις γλώσσες και από όλες τις γλώσσες. Η κυρία Γέγελα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα να σας ενημερώσω έτσι, σύντομα για την ε, τρέχουσα κατάσταση του τριμερούς διαλόγου για την οδηγία για τα πειραματόζωα. Εδώ και ένα μισή χρόνο ασχολούμαστε με αυτό το θέμα εντατικά και χαίρομαι για το ότι στις 7 Απριλίου αφού στις 7 ε, Δεκεμβρίου είχαμε το πρώτο τμήμα του συμβασμού, τώρα ολοκληρώσαμε και το δεύτερο μέρος. Στον τελευταίο αυτόν ε, τριμερή διάλογο θέμα ε, είναι αυτό το οποίο λέγαμε παλιά επιτροπολογία και αυτό το οποίο σήμερα λέμε πράξεις κάτω εξουσιοδότηση, οπότε είμαστε στο πλαίσιο της Λισαβόνας για να βρούμε μια συμβιβαστική λύση που θα ενισχύει εμάς, το Κοινοβούλιο. Και νομίζω ότι τα καταφέραμε αρκετά καλά. Όμως θα ήθελα αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμότατα όλους όσους συνεργάστηκαν τον 1,5 αυτών χρόνων. Να ευχαριστήσω τους ε, συνεργάτες των διαφόρων υπηρεσιών εδώ στην Επιτροπή, κυρίως τον Πάτρικ, να ευχαριστήσω τους συνεργάτες και των ομάδων, όλων των πολιτικών ε, ομάδων και εδώ πέρα είχαμε στενή συνεργασία, όλους τους κοιόδης συγητές ε, και συγγητρίους στην Κομισιόν, τη Σουηδική και την Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου. Η οδηγία, όπως έχει αυτή τη στιγμή για την προστασία πειραματόζων είναι από το 1986 και στόχο έχει να επιτύχει ίδιες συνθήκες πλαίσιο για την προστασία των πειραματόζων σε όλο αυτόν τον κλάδο και να είναι βέβαια δεσμευτική πανευρωπαϊκά. Καταφέραμε λοιπόν και στόχο έχει να κατατάξουμε τον πόνο τον οποίο υποφέρουν αυτά τα ζώα. Οπότε πειράματα σε ζώα δεν θα πρέπει να γίνονται χωρίς πρώτερη αδειοδότηση των αρμοδίων αρχών. Με άλλα λόγια, κανένα έργο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εάν δεν έχει υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα της αξιολόγησής του εκ των προτέρων οι ηθικές σκέψεις και αξιολογήσεις θα πρέπει να αφορούν το πόσο συμβιβάζεται αυτό το πείραμα με τις απαιτήσει τις δικές μας απαιτήσει δηλαδή της ε, μείωσης ε, της αποφυγής και της βελτίωσης κατάστασης των ζώων και επίσης θα υπάρξει και μια αναδρομική αξιολόγηση, κάτι το οποίο είναι καινούριο. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να συστήσει μια Εθνική Επιτροπή Προστασίας των Ζώων και Ηθικής που θα συμπεριλαμβάνει βέβαια και τις αρμόδιες αρχές ε, και τα φόρα προστασία των ζώων και θα πρέπει να υπάρξει επίσης ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Επίσης θα πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικέ ε, των πειραμάτων σε ζώα εφόσον είναι νομικά αναγνωρισμένες και θα πρέπει να περιοριστεί σε ένα ελάχιστο αριθμό των χρησιμοποιούμενων ζώων. Επίσης τα κράτη ζώα υποχρεώνονται να δουν ε, τα της ε, διατροφής και διαβίωσης ε, των ζώων και περιορισμού των αριθμών τους έτσι ώστε για να μπορέσει να περιοριστεί ο πόνος αυτών των ζώων. Έχουμε λοιπόν αυτό τον, τον στόχο, μείωση, αντικατάσταση και μια, έτσι, των μεθόδων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις όπως και στην πρώτη ανάγνωση 5 Μαΐου 2009 διευκρίνησε πως πρέπει να γίνουν περισσότερα για να φτάσουμε στον στόχο της πλήρους αντικατάστασης των ζώων από τα πειράματα. Αυτό είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος μας, αλλά συμφωνούμε πως ακόμα σήμερα δεν είμαστε στη θέση να αντικαταστήσουμε τελείως τα ζώα. Μετά λοιπόν από 1,5 έτος εντατικών συζητήσεων στο Κοινοβούλιο και μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιών, καταφέραμε να επιτύχουμε μια λεπτή ισορροπία μεταξύ έρευνας και προστασίας των ζώων, που βεβαίως προστατεύει και τα συμφέροντα των επιχειρήσεων που κάνουν έρευνα και βεβαίως έχουν στόχο την ανθρώπινη υγεία, αλλά θα έχει στόχο βεβαίω και την υψηλότερη δυνατή προστασία των ζώων με το να δώσουμε το παγκόσμιο παράδειγμα σε αυτές τις ε, προδιαγραφές χωρίς όμως να διακινδυνεύσει η έρευνα στην Ευρώπη. Όλοι οι σκιώδεις εισηγητές συμφώνησαν σε αυτή τη συμβαστική λύση. Γι' αυτό σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε να αποστείλετε μια επιστολή εξ ονόματος της Επιτροπής μας στην Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου έτσι ώστε επισήμως να συμφωνήσουμε και εμείς. Για τα περαιτέρω θα έπρεπε ίσως να ξέρετε πως η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου ασχολείται πάρα πολύ σοβαρά με αυτό το θέμα. Στο δε συμβούλιο τα ψάχνουν λέξη-λέξη, ελέγχουν αυτή τη στιγμή τις παραπομπές ε, στην ανάλογη νομοθεσία και αν είναι σωστά, ε, σωστή η νομική γλώσσα. Και μετά θα επανυποβληθεί σε εμάς αυτή η έκθεση και θα μπορέσουμε να την συζητήσουμε σε μια συνεδρίαση δική μας έτσι ώστε να έχουμε μια δεύτερη ανάγνωση του Κοινοβουλίου και ελπίζουμε ακόμα επί Ισπανικής Προεδρίας αλλά ίσως μάλλον τον Σεπτέμβριο να ολοκληρώσουμε. Αυτό εξαρτάται από το χρονοδιάγραμμα και τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν και σας παρακαλώ να τις στηρίσουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Ελίζαμπεθ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική σου εργασία. Τώρα θα ξεκινήσουμε με την παρουσίαση της μελέτης. Η συνεδρία να μεταδίδεται μέσω web stream και θα ξεκινήσουμε με την παρουσίαση της μελέτης σχετικά με την υλοποίηση του ελέγχου της υγείας της κοινή ε, γεωργικής πολιτικής στα κράτη-μέλη, ειδικότερα σε συνάρτηση με τα νέα άρθρα 6869 του κανονισμού αριθμός 73-2009. Καλώς ορίζω τους κυρίους Έμον Μπίτς ε, και τον ε, κύριο Γουίμερ, που είναι και οι συντάκτες της μελέτης και δίνω το λόγο στον κύριο Πίτς για να παρουσιάσει τη μελέτη. Θα συνεχίσουμε με μια σύντομη συζήτηση σχετικά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ο Ήμον Πίτς και παρουσίασα αυτή την μελέτη, παρουσιάζω αυτή τη μελέτη εξ ονόματος της ΜΕΤΙΣ. Αφορά την εφαρμογή του check-up στα κράτη-μέλη. Τη ζήτησε το Κοινοβούλιο, οπότε προφανώς σας ενδιαφέρουν οι λεπτομέρειες του πώς ε, εφαρμόζεται αυτή η αλλαγή πολιτικής στην πράξη. Αυτό το οποίο μας ζητήσατε δηλαδή να δούμε. Εάν δείτε τώρα αυτή την παρουσίαση, θα δείτε αυτό που θα σας πω εγώ, δηλαδή θα συνοψίσω τους στόχους, το υπόβαθρο του κανονισμού και μετά θα δούμε το πώς εφαρμόζεται ο κανονισμός και μετά θα έχουμε κάποιες παρατηρήσεις για τα ευρήματα. Τα ευρήματα ε, είναι βεβαίως το κομμάτι της εφαρμογής. Αυτά είναι τα, τα νέα μας και μετά θα δούμε κάποια σχόλια για τα ευρήματά μας. Λοιπόν, υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα. Έχουμε την αποσύνδεση των πληρωμών, υπάρχει επιλογή του μοντέλου πληρωμής και ένα ακόμα ζήτημα, οι εθνικές επιδοτήσεις. Αυτό σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, καθώς στον τίτλο της μελέτης υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά στα άρθρα 68 και 69. Όταν μας ζητήσατε την μελέτη φαίνεται πως σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό, οπότε θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας. Οπότε, ποιοι ήταν οι στόχοι της ε, μελέτης, τι θέλατε να εξακριβώσουμε. Πρώτος στόχος είναι να ξέρετε από νωρίς το πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο της ΚΑΠ όταν θα εφαρμοστούν πλήρως οι αλλαγές. Ετέθησε ισχύ το check-up πριν από ένα έτος, οπότε είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Βεβαίως υπάρχουν κάποια σημάδια και εσείς θέλατε κάποια ένδειξη για το τι συμβαίνει. Ειδικά δεδομένου του ότι αλλού γίνονται διαπραγματεύσεις, ακόμα και αυτή τη στιγμή μιλάμε για αλλαγή της πολιτικής, οπότε σας ενδιαφέρει το τι συμβαίνει στις αλλαγές που είχαν συμφωνηθεί πριν από 18 μήνες. Οπότε δεύτερος στόχος είναι να δούμε τις επιλογές των κρατών μελών. Αυτό το οποίο προέβλεπε λοιπόν ο κανονισμός ήταν ε, κάποιες επιλογές, δηλαδή υπήρχε μία δυνατότητα ανεξάρτητης κίνησης των κρατών μελών και εμείς μετά είδαμε ποιες ήταν αυτές οι επιλογές και πως κρατη κράτη-μέλη επέλεξαν τη μία ή την άλλη λύση και μετά κάποια ανάλυση με βάση τις πληροφορίες που λάβαμε. Η μέθοδος ήταν έρευνα και ερωτηματολόγιο. Δεν έχουμε λάβει ακόμα όλα τα ερωτηματολόγια. Ελπίζουμε να γίνει αυτό σε μερικές εβδομάδες, αλλά είχαμε κάποια κενά σε ένα ιδιαίτερο ζήτημα όπου δεν γνωρίζουμε τις προθέσεις των μελών και θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Τώρα, η βασική νομοθεσία εδώ πέρα είναι ο κανονισμός 73 του 2009 που αφορά την ενιαία πληρωμή αν εκμετάλλευση. Εφαρμόζει κάποιες πτυχές του check-up. Το check-up το οποίο περιείχε μεγάλες αποφάσεις ε, κατήργησε την αγρανάπαυση ε, και Δώσε επίσης μεγαλύτερο βάρος στην διάρθρωση, αλλά όλα αυτά τα πράγματα δεν περιέχονται στο 73-2009. Πρόκειται για ένα πολύ τεχνικό κανονισμό και αφορούσε αυτά τα τεχνικά ζητήματα, την αποσύνδεση δηλαδή, την επιλογή συστήματος πληρωμής και τις εθνικές επιδοτήσεις που αποτελούν τμήμα της ενιαίας επεπληρωμής ανά εκμετάλλευση. Αυτά τα τρία τεχνικά ζητήματα λοιπόν προέκυψαν από τον κανονισμό. Πρώτα απ' όλα αποσύνδεση. Ο κανονισμός όριζε το 2012 ως προθεσμία για τις συνδεδεμένες με την παραγωγή επιδοτήσεις. Πλην βεβαίως τη λαζόνα γελάδων, προβάτων και κάποιων επεξεργασμένων ε, οπροκυπευτικών που θα μπορούσε να συνεχίσει μέχρι και μετά το 2012. Τι συνέβη. Εν ολίγης θα επιτευχθεί ο στόχος. Κάποιες χώρες μάλιστα ήδη τον εφαρμόζουν πριν από την προθεσμία. Πέρσι υπολόγισε ένα αξιωματούχος κομισιόν πως 87% της άμεσης στήριξης ήταν ήδη αποσυνδεδεμένη. Και άρα μέχρι το 2012 θα έχουμε φτάσει γύρω στο 99%. Θα υπάρχει ακόμα ένα μικρό ποσοστό επιδοτήσεων συνδεδεμένων, αλλά το ποσοστό συνολικών επιδοτήσεων θα είναι αμεληταίο, το συνδεδεμένων. Κάτι το οποίο θα φανεί αργότερα. Υπάρχουν νέες συνδεδεμένες επιδοτήσεις που εισάγονται παράλληλα. Δεν έχουν μεγάλη σημασία, αλλά εάν μιλάμε για αποσύνδεση, πρέπει να γνωρίζουμε πως παράλληλα με την αποσύνδεση επιτρέψαμε κάποιες νέες συνδεδεμένες επιδοτήσεις. Οπότε, τι γίνεται με την αποσύνδεση. Δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εδώ πέρα. Ο στόχος θα επιτευχθεί και μάλιστα και πριν την προθεσμία. Τώρα, το άρθρο 63 που συνδέεται με τη διαδικασία αποσύνδεσης και δίνει μια νέα επιλογή στα κράτη-μέλη. Κανονικά, όταν γίνεται η αποσύνδεση, η πληρωμή ενσωματώνονταν στην ενιαία πληρωμή αναεκμετάλλευση. Αυτό αναμέναμε. Στο άρθρο 63 όμως είχαμε μια νέα διάταξη η οποία επέτρεπε στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα της αποσύνδεσης για να υποστηρίξουν καλλιέργειες, ε, γεωργικές δραστηριότητες που δεν σχετίζονταν με τη συνδεδεμένη πληρωμή. Η Γαλλία το χρησιμοποίησε σε μεγάλο βαθμό όταν αποσύνδεσαν τις ε, αρωτρέες καλλιέργειες που ήταν αρκετά μεγάλες πληρωμές και τις ε, εγώ προβάτων και σφαγής βοηδών, τα κονδύλια αυτά πήγαν σε διαφορετικές ομάδες αγροτών π.χ. βοσκοτόπων και των αναλόγων καλλιεργειών. Οπότε υπήρχε μια μεγάλη μεταφορά επιδοτήσεων ε, από τον ε, τομέα των αρωτέρων καλλιεργειών, στον τομέα των ε, βοσκοτόπων και ζωοτροφών. Όπως είπα, καμία άλλη χώρα δεν το έκανε σε τόσο μεγάλη κλίμακα, αλλά και η Γερμανία και η Φιλανδία σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την επιλογή σε μικρότερη κλίμακα μέχρι το 2012. Περνάμε τώρα στο δεύτερο ζήτημα το οποίο αφορά το μοντέλο των πληρωμών. Το 2003 είχαμε προβλέψει μια επιλογή του μοντέλου πληρωμών. Σε όλες τις φάσεις, λοιπόν, είχαμε ένα μοντέλο στο οποίο θα είχαμε την ίδια πληρωμή με πιθανές ε, περιφερειακές παραλλαγές. Αλλά υπήρχε, βεβαίως θα θέλαμε να υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο, αλλά υπήρχαν επιλογές μπορούσαν να κάνουν τα κρατημέλη. Λοιπόν, τα παλαια κρατημέλη επέλεξαν ένα ιστορικό μοντέλο και υπήρχε ένα υβριδικό, αν θέλετε, μοντέλο μεταξύ των ιστορικών δικαιωμάτων και του ε, νέου μοντέλου. Τα νέα κρατημέλη μπορούσαν βέβαια να επιλέξουν κάτι απλούστερο. Ο νέος κανονισμός του 2009 συνέχισε σε αυτή την κατεύθυνση και αυτές οι επιλογές θα μπορούν να διατηρηθούν μέχρι το 2012. Οπότε στα παλιά κρατημέλη είναι ακόμα δυνατόν να διατηρηθεί το ιστορικό μοντέλο. Στα νέα κρατημέλη είναι δυνατόν να διατηρηθεί το μοντέλο SAPS μέχρι να αλλάξει αυτή η το 2012. Τι σημαίνει λοιπόν, τι έχει αλλάξει είδαμε από τα 27 καρτιμέλη πόσες χώρες ακολουθούν το προτιμόμενο μοντέλο. Μόνο δύο λοιπόν είναι αυτές, η Σλοβενία και η Μάλτα. Τρεις χώρες σκοπεύουν να εφαρμόσουν αυτό το προτιμόμενο μοντέλο μέχρι το 2012. Η Ουγγαρία, η Λετωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ηνωμένο Βασίλειο μόνο στην Αγγλία. Η δε Γερμανία σκοπεύει να το εφαρμόσει το 2013. Ανέφερα πριν πως η μελέτη δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα ερωτηματολόγια δεν απαντήθηκαν από όλες τις χώρες, οπότε μάλλον υπάρχουν και κάποιες άλλες χώρες που σκοπεύουν να εφαρμόσουν το σύστημα αυτό της ίδιας πληρωμής μέχρι το 2012. Όπως είπα δεν έχουμε ακόμα λάβει όλα τα ερωτηματολόγια. Από τα 15 κράτη-μέλη, ε, τα παλιά 15 κράτη, λειτουργούν με το παλιό σύστημα και έξι με υβριδικό σύστημα. Το Ρωμανό Βασίλειο με το δικό του τρόπο. Έχει και τα δύο συστήματα. Οχτώ από τα δύο συστήματα χρησιμοποιούν ακόμα το SAFS. Και δεν υπάρχουν σχέδια μετά από το ερευνητολόγιο. Διαπιστώσαμε σε πολλές χώρες δεν υπάρχει καμία πρόθεση να εισαχθεί το προτιμόμενο σύστημα μέχρι το 2012. Δεν υπάρχουν λοιπόν τέτοιες προβλέψεις της σε πολλές χώρες. Έχουμε εδώ πέρα μια χτυπητή αντίθεση για το θέμα αυτό, όπως και για το θέμα της αποσύνδεσης. Για την αποσύνδεση γίνονται πράγματα με μεγάλη ταχύτητα, εδώ υπάρχει χελωνοδρομία. Μία παράπλευρη υπόθεση σε σχέση με τα νέα κράτη-μέλη τώρα. Είναι το θέμα των συμπληρωματικών εθνικών άμεσων πληρωμών τα νέα μέλη είχαν τη δυνατότητα να προσθέτουν, να συμπληρώνουν με εθνικούς πόρους τις πληρωμές αυτές με την, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου μέχρι το 2012 για τις 10 νέες χώρες και για το 2016 για τη Ρουμανία αλλά και τη Βουλγαρία. Αυτή η επιλογή λοιπόν υλοποιήθηκε στις περισσότερες από τις νέες χώρες μέλη. Πέραν επομένως των ε, επιδοτήσεων που προέρχονται από τα ευρωπαϊκά ταμεία υπάρχουν και οι εθνικές επιδοτήσεις οι οποίες δίνονται στις χώρες αυτές. Κάποιες από αυτές τις επιδοτήσεις είναι συνδεδεμένες. Αλλά γενικά είναι μικρός ο βαθμός σύνδεσης και αφορά <clears throat> γενικά δύο τομείς αυτή η σύνδεση. Αυτές οι πληρωμές θα μειωθούν καθώς πλησιάζει η μεταβατική περίοδο και αυξάνονται αντίστοιχα ή ευρωπαϊκού χαρακτήρα πληρωμές θα καταργηθούν σταδιακά οι εθνικές πληρωμές με το 2012 ή 2016 αντίστοιχα. Ένα τρίτο θέμα το οποίο ατενίζουμε είναι οι εθνικά επινοημένες επιδοτήσεις, αν θέλετε, άρθρα 68 και 69. Στην νομοθεσία του 2003 προβλεπόταν να υπάρξει ειδική υποστήριξη στην ε, γεωργία που επιτρέπει το σημείο της Ενίας πληρωμής. Τα κράτη-μέλη μπορούσαν να φτάσουν ένα 10% του εθνικού ε, συστήματος, του εθνικού, μάλλον της εθνικής οροφής. Επίσης, ε, οι στόχοι αυτής της επιδότησης θα έπρεπε να είναι να υποστηρίξουν την ποιότητα ή την προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά με τον νέο κανονισμό του 2009 έχουν διευρυνθεί οι στόχοι οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετηθούν και μειώνεται και η γραφειοκρατία. Η κύρια αλλαγή είναι ότι οι επιδοτήσεις επιτρέπονται τώρα για να υποστηρίξουν οικονομικά τροτές περιοχές ή είδη γεωργίας στον τομέα της ε, παραγωγής βοήου κρέατος, γαλακτοκομικών, προβίου κρέατος και επίσης την καλλιέργεια ορίζης. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα να υποστηρίξουμε οικονομικά εύθραυστες δραστηριότητες ως τμήμα της ενιαίας πληρωμή. με αυτόν τον τρόπο επανερχόμαστε σε κάποιο βαθμό περιορισμένο στην ενιαία, ε, στις ενιαίες πληρωμές. Τι γίνεται τώρα στην πραγματικότητα. Τα άρθρα 68 και 69 εφαρμόζονται το 2010 σε 22 κράτη-μέλη, ενώ ήταν μόνο 8 το 2007 βάσει του παλαιού κανονισμού. Υπάρχει λοιπόν μια ουσιαστική αλλαγή σε επίπεδο δραστηριοτήτων. 14 κράτη-μέλη έχουν προγράμματα στο γαλακτοκομικό τομέα για να τον υποστηρίξουν. Βλέπετε μπροστά σας να λέει το γράφημα 7 στα εγωπρόβατα. Όχι, είναι 8 γιατί και η ελλαδική κυβέρνηση εισήγαγε την προηγούμενη εβδομάδα ένα νέο ε, πρόγραμμα υποστήριξης για τα αρνιά και τα τραγιά. Τα κράτη-μέλη λοιπόν που έχουν τέτοιο είδους υποστήριξης είναι 8 και τρία που αφορούν το βόλιο κρέα. Ποιε είναι οι άλλε τώρα δυνατότητε, Προγράμματα για την ασφάλεια των ε, καλλιεργειών ή των ζωικών ε, εκτροφών. Τέσσερα κατημέλη ζητήσανε να έχουν τέτοια προγράμματα. Μία ακόμα περαιτέρω επιπλέον επιλογή είναι να υπάρχει προστασία εναντίον των ε, ασθενειών των ζώων και εναντίον των ε, ασθενειών των φυτικών καλλιεργιών. Μόνο για τη Γαλλία υπάρχει αυτή, υπήρξε αυτή η επιλογή το 2011. Τα, προβλήματα, τα προγράμματα ποιότητος και τα προβλήματα περιβάλλοντος τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν <clears throat> συνεχίζουν. Δεν εφαρμόζονται βέβαια στην ίδια κλίμακα. Επομένως τα κράτη-μέλη σε μεγάλο βαθμό έχουν αντικαταστήσει με νέα προγράμματα τα παλιά τέτοια προγράμματα. Είπαμε ότι μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει μέχρι 10% τη οροφή. Πόσες χώρε το πράττουν αυτό όμως. Και βλέπετε στο επόμενο γράφημα, στον επόμενο πίνακα, ότι υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία. Υπάρχουν πέντε χώρε οι οποίες εφέτος έχουν σαν στόχο να δαπανίσουν πάνω από 7,5% του εθνικού ανώτατου όριου, τη Εθνική οροφή Και έχουν ευρεία γεωγραφική κατανομή. Φιλανδία, Ιταλία, Ουγγαρία, Ελλάδα και Σλοβενία. Ακολουθεί μια ομάδα χωρών 4,8 με 5,7 περίπου το μισό, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Τσεχική Δημοκρατία και Λετωνία. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν πέντε χώρες που δεν χρησιμοποιούν καθόλου αυτό το σύστημα. Βέβαια, η πλήρης έκθεση που έχετε δείχνει ότι μάλλον υπάρχει κάποιο πρόγραμμα στη Σκωτία, δεν είναι απόλυτα σωστό να πούμε μηδέν χρηματοδότηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία και η Γερμανία κάτω από 1% και υπάρχει και μια ομάδα άλλων χωρών που δαπανούν μεταξύ 1 και 2%. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη πολυπικιλία σε σχέση με την υιοθέτηση από την πλευρά των κρατών μελών για τα προγράμματα αυτά. Ορισμένε χρησιμοποίησαν την δυνατότητα για να δαπανίσουν μέχρι και 10% τη οροφή σε προγράμματα που έχουν αναπτύξει οι ίδιε αυτέ χώρε. Άλλε όμω δαπανούν ελάχιστα ποσά. Τώρα, κανονισμός προβλέπει ότι μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση είτε από εξοικονομήσεις σε άλλα κονδύλια ή σε μια γραμμική μείωση της ενίας τρεματικής ενίσχυσης ή σε ένα συνδυασμό και των δύο. Η Γαλλία δέχτηκε και η Ιταλία διαλέξαν να μειώσουν την ενιαία πληρωμή κατά 4,5 και μέχρι 3,8 στην περίπτωση Ιταλία. Ορισμένα κρατημέρια χρησιμοποιούν μονάχα την οδό των εξοικονομήσεων και γι' αυτό έχουν τόσο χαμηλό ποσό χρησιμοποίηση σε σχέση με τα εθνικά κατόφλια, οι χώρε που είναι 1 με 2% ή πιο κάτω. Σίγουρα οι χώρες αυτές δεν μειώνουν την ενιαία πληρωμή. Η πιο κατω σιγουρα οι χώρε αυτέ δεν εικόνα για τον αντίκτυπο του άρθρου, των άρθρων 68 και 69 είναι ότι το 2010 υπολογίζουμε ότι η συνολική εκταμείευση για τα προγράμματα αυτά θα είναι περίπου 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ήταν μόνο 4,25 εκατομμύρια το 2009. Δηλαδή μια, ένα, μια διαδικασία τετραπλασιασμού. Και συνολικά είναι 4% του εθνικού, των εθνικών οροφών. Παρατηρήσεις τώρα, επειδή ίσως δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Η αποσύνδεση λοιπόν έχει ξεπεράσει αυτό το οποίο προβλεπόταν το 2003. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν μεγάλη επιλογή για την εφαρμογή της αποσύνδεσης. Απλώς να τη διαλέξουν, να την εφαρμόσουν πλήρως ή όχι η ταχύτητα με την οποία εφαρμόστηκε η αποσύνδεση θα έπρεπε να βελτιώσει τη διαπραγματευτική θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνές συζητήσεις και συμφωνίες για το εμπόριο, αλλά έχουν εισαχθεί και νέε συνδεδεμένε επιδοτήσει σε μέτρα του άρθρου 68 και σε συμπληρωματικέ αντισταθμιστικέ εθνικέ πληρωμέ. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το γενικό, τη γενική πορεία προ την αποσύνδεση. Για τα συστήματα πληρωμών έχουμε μια κατάσταση η οποία δεν αντανακλά την προτιμητέα κατάσταση υπήρξε μια ελάχιστη κίνηση για το σύστημα καταποκοπή και πρέπει να ρωτήσουμε γιατί. Εδώ επί επίπεδου οικοτολογίας μονάχα μπορούμε να απαντήσουμε. <clears throat> Καταρχήν, το 2012 ως στόχος είναι κάπως μακρόπνος. Γιατί να κάνουμε κάτι το 2010 και το 2011. Η γραφειοκρατική λοιπόν στάση είναι συνήθως να τα εφαρμόσουμε όλα τελευταία στιγμή και όχι να τα κάνουμε πρωτού χρειάζεται. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που θα αλλάξει η πολιτική. Και πολλοί σκέφτονται γιατί να αλλάξουμε μια πολιτική όταν <clears throat> ούτως ή άλλως θα την ξαναλλάξουμε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Και πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο δεν γίνονται πολλά πράγματα για την εφαρμογή του νέου συστήματος. Λένε πολλοί ότι περνάμε τώρα στη διαδικασία διαπραγμάτευσης ενός νέου συστήματος γιατί να σκοτιζόμαστε να εφαρμόσουμε μια αλλαγή την οποία μετά θα πρέπει να την ανατρέψουμε και πάλι το 2013. Και επίσης υπάρχει ένας αριθμός χωρών που θα προτιμούσαν να διατηρήσουν τις ιστορικές βάσεις πληρωμών. Να κρατήσουν λοιπόν την ιστορική αυτή βάση. Τώρα αν θα μπορούν να το πετύχουν αυτό ή όχι σε διαπραγματεύσει, αυτό παραμένει να το δούμε. Αλλά αν είσαστε υπουργό ο οποίο προτιμάει να διατηρήσει μια ιστορική βάση πληρωμών, δεν θα δεχτείτε να κάνετε γρήγορες αλλαγές. Για τις εθνικές επιδοτήσεις τώρα. Η χρήση του άρθρου 68 ήταν πολύ πιο διαδεδομένη από ό,τι στον κανονισμό του 2003 και ιδίω είναι δημοφιλή τα μέτρα υποστήριξη του γαλακτοκομικού τομέα. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από την πλευρά των κρατών μελών σε σχέση με την χρησιμοποίηση ή όχι του μέχρι 10% των εθνικών ε, οροφών. Και νομίζω ότι μπορώ να κλείσω εδώ Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βοήθεια που μας έδωσε και τους εθνικούς εμπειρογνώμονες, τους αξιωματούχους από τα κράτη-μέλη. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς για την προσοχή σας και είμαι έτοιμος να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Thank you. spoke about... Όταν μιλήσατε για την <clears throat> χρησιμοποίηση των εξοικονομήσεων για το άρθρο 68-69. <clears throat> Τι ακριβώς είχατε στο μυαλό σας. Ο κανονισμός το προβλέπει αυτό. Ότι έχει τεθεί ένα εθνικό, μια εθνική οροφή και αν υπάρχουν ποσά τα οποία βρίσκονται μέσα στο εθνικό όριο αυτό που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί βάση των συγκεκριμένων ε, άλλων διατάξεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα ποσά βάσει του άρθρου 68 και 69. Λοιπόν, μισό λεπτό κύριε Πίτς ε, πριν, ε, πριν, πριν απαντήστε, γιατί πρέπει να μαζέψουμε πολλές ερωτήσεις. Ο Άλμπερτ και μετά ο Λουίς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την παρουσίαση που μας έχει κάνει. Εγώ, σαν συντονιστής, ενδιαφέρομαι για την ε, έκθεση αυτή. Δεν θέλω τώρα να ψέξω τους εμπειρογνώμονες οι οποίοι έχουν κάνει αυτή την έκθεση, αλλά έχει νόημα να υπάρχει μια τέτοια έκθεση από εμπειρογνώμονες και όχι από την ίδια την Κομισιόν. Νομίζω ότι θα έπρεπε η Κομισιόν να χρησιμοποιήσει τις ε, εκθέσεις των εθνικών κρατών και να τις ε, συμπηλήσει για να τις φέρει ενώπιον της Επιτροπής μας. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να δίνουμε ποσά για να εκπονηθεί μια τέτοια ε, έκθεση και η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών ίσως δεν θα είναι πολύ ευχαριστημένη με όλα αυτά τα θέματα για την αποσύνδεση τώρα. Υπάρχει στη Γερμανία αυτός ο χρόνος μετάβασης τριών-τεσσάρων ετών για να υπάρξει πλήρης εφαρμογή της ε, αποσύνδεσης. Αλλά υπάρχουν μέσα στο πλαίσιο αυτό ορισμένοι γεωργοί σε μειονεκτικές περιοχές οι οποίοι θα είναι κατά κάποιο τρόπο οι χαμένοι αυτής της υπόθεσης και υπάρχουν άλλοι που βρίσκονται σε πιο θετική στάση. Αλλά νομίζω ότι η χρήση αποκλειστικά και μόνο της διαδικασίας αποσύνδεσης δεν επιλύει όλα τα προβλήματα. Αντίθετα, για ορισμένε περιοχές θα πρέπει να συζητήσουμε αν θα πρέπει να εφαρμοστεί η αποσύνδεση όπως προβλεπόταν, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που θα αντιμετωπιστούν από αυτές τις περιοχές όπου υπάρχουν γεωργοί οι οποίοι κινδυνεύουν πραγματικά να μην μπορούν να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους. Όπως είπε λοιπόν και ο, και ο αρμόδιος εμπειρογνώμων, δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο αυτό το οποίο μας είπε, ότι υπάρχουν πολλοί υπουργοί σε κράτη-μέλη οι οποίοι δεν θέλουν να εφαρμόσουν αυτό το σύστημα γιατί σκέφτονται τα ιστορικά δεδομένα. Ο Ευχαριστώ Άλμπερτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την παρουσίαση που έγινε από τον κύριο Πιτ. Γιατί όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τη γνώση της πραγματικότητας και ιδίως της πρόσφατης πραγματικότητας είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για μας τους ε, νομοθέτες οι οποίοι πρέπει να εμπλακούμε σε μια πολύπλοκη διαδικασία για το μέλλον. Επομένως, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η μελέτη η οποία παρουσιάστηκε ενώπιον. Και φυσικά αυτή η μελέτη μας αναγκάζει να σκεφτούμε καλύτερα έναντι της ε, θέλησης που έχουμε όλοι να έχουμε μια πολιτική όσο το δυνατόν πιο εναρμονισμένη για να είναι ισοδίκαια, ενώ συγχρόνως διαπιστώνουμε ότι όταν δίνουμε στα κράτη-μέλη κάποια ευελιξία, κάποια δυνατότητα προαιρετικών μέτρων, τότε το αποτέλεσμα είναι ότι πολύ γρήγορα αυτή η πολιτική πάβει να έχει τον ενιαίο και κοινοτικό χαρακτήρα της. Είναι σαφές ότι αυτή η, μετάφαση, αυτή η μετάβαση από την παλιά κοινή αγροτική πολιτική προς τη νέα αγροτική πολιτική του 2013 και επέκεινα προϋποθέτει μια τέτοια άσκηση ευελιξίας. Συγχρόνως όμως θα πρέπει να δούμε τι μας λένε οι μελέτες εφαρμογής αυτών των πολιτικών για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια πιο ισοδίκαια πολιτική στο μέλλον, χωρίς φυσικά να απολεστεί ο κοινότικό χαρακτήρας της. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που συνέταξαν αυτή την έκθεση και τονίζω ότι έχει μεγάλη σημασία και ωφέλεια για όλους μας. Ο πρόεδρος ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα τα στοιχεία που δόθηκαν σχετικά με την εφαρμογή ή μη εφαρμογή των άρθρων. Μιλήσαμε πολύ για αυτή τη δυνατό, τις δυνατότητες και πολλά κράτη-μέλη είδαμε δεν εκμεταλλεύονται απόλυτα τις δυνατότητες που προσφέρουν αυτά τα άρθρα. Και αυτό είναι και το αντικείμενο της ανάλυσης που έγινε, δηλαδή γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί υπάρχει τέτοια διαφορά ερμηνείας και εφαρμογή των άρθρων αυτών στα κράτη-μέλη. Ερώτηση. Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία απευθύνθηκαν προς την Κομισιόν για μία υποστήριξη και δεν τους δόθηκε. Αν δεν υπάρχουν άλλοι που θέλουν το λόγο, μαγκίνες. Μερσή κύριε Πρόεδρε. Και θέλω ευχαριστώ τον Ιαμον Πίτς για τη μελέτη μας παρουσίασε. Νομίζω ότι είναι απόλυτα ορθό να πούμε ότι αυτά μας παρουσιάζουν την κατάσταση στα κρατη θα ήθελα ο κύριος Πίτς να κάνει κάποια σχόλια, αν υπάρχει κάποια ανάλυση για τον απόϊχο αυτών των μέτρων και τα, τις επιπτώσεις, δεν ξέρω αν είναι πρόωρο να γίνει κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να μας δώσει και περισσότερα στοιχεία σε σχέση με την πληροφόρηση που μας είπε ότι υπάρχει λίγη κίνηση προς ένα σύστημα κατά αποκοπήν πέραν αυτών που παρουσιάστηκαν στα, στις, στα γραφήματα σχημάτισε κάποια εντύπωση ο κ. Σπίτς και οι συνεργάτες του από τα ερωτηματολόγια τα οποία συνέλεξη, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Και τέλος το θέμα της δικαιοσύνης μέσα σε εισαγωγικά του συστήματος. Είναι κάτι για το οποίο ακούμε πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ λίγη σύμφωνη για το τι σημαίνει ένα ισοδίκαιο σύστημα. Ίσως είναι άδικο το ερώτημα αυτό προς ένα ερευνητή αλλά θα μας βοηθούσε πολύ αν μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες ιδέες, κάποια στοιχεία για το τι αποτελεί ένα δίκαιο σύστημα. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, ακούγον τις λεπτομέρειες του συστήματος αυτού αυτό ενισχύει την εντύπωση που έχω για την πολυπλοκότητα αυτού που στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν μια απλή ιδέα. Το άρθρο 68, το άρθρο 69 ήταν στην αρχή απλές ιδέες. Αλλά ο τρόπο με τον οποίο ερμηνεύτηκε και εφαρμόστηκε στα κράτη-μέλη φαίνεται ότι είναι δεδαλώδε και πολύπλοκο. σω είναι χρήσιμο να έχουμε την ευελιξία, αλλά θα ήθελα να ξέρω και την άποψη του κ. Πιτ για αυτά. Ε, ο Ζωζέ ζήτησε το λόγο. Καλώς ορίζω και τον Επίτροπό μας στο μεταξύ, ο Ζωζέ Μποβέ. Μία παρατήρηση σύντομη, γιατί δεν αναφέρθηκε καθόλου στις εξηγήσεις που μας δόθηκαν. Αν περάσουμε σε αυτή τη μορφή υποστήριξης, τότε βρισκόμαστε σαφέστατα στα πλαίσια ε, των όσων επιβάλλει η ΠΟΕ και έχουμε μεταφορές είτε στο πράσινο κουτί είτε στο πορτοκαλί κουτί και τελικά επικαλύπτουμε την πραγματικότητα. Δεν πρόκειται εδώ δηλαδή για καλή θέληση των κρατών μελών αλλά πρόκειται για μια εσωτερική ρύθμιση της αγοράς. Και ποια είναι μια σημαντική επίπτωση αυτής της νομοθεσίας στο βαθμό που ξεχωρίστηκαν οι, οι ενισχύσεις είδαμε να πέφτουν οι τιμές των αγροτικών προϊόντων και έμεσα δηλαδή όλο αυτό λειτουργήσε σαν ενίσχυση είτε στις μεγαλοβιομηχανίες είτε στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Έχουμε μια μεταφορά λοιπόν η οποία γίνεται τεχνητά από τον ε, καταναλωτή είτε από τον φορολογούμενο. Δηλαδή και οι δύο λειτουργούν ως αγελάδες για άρμεγμα. Και αυτό γιατί, γιατί ακολουθήσαμε τους ε, κανόνες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου και ακολουθήσαμε δηλαδή ότι μας επέβαλαν οι διάφορες ε, συμφωνίες που υπογράψαμε. Αν δεν θέλει κανένας άλλος το λόγο να μιλήσει ο κύριος Πίτς, έχει τρία λεπτά στη διάθεσή του. Ε, ε, ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Κάποια από τα σχόλια ήταν περισσότερα σχόλια και όχι ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες από τις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ένας βουλευτής ρώτησε γιατί δεν εφαρμόζονταν το άρθρο 68 σε κάποια κράτη-μέλη. Δεν νομίζω πως είναι σωστή αυτή η οπτική. Υπήρχε μια επιλογή που είχαν τα κρατη Εάν το έκαναν αυτό, ε, γενικά κάτι τέτοιο σημαίνει πως θα περικόψουν το επίπεδο της ε, ενιαίας πληρωμής όλων για να ενισχύσουν μια συγκεκριμένη ομάδα αγροτών. Ξέρω πως η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου, παραδείγματο χάρη, είναι πως δεν θένε να μειώσουν την ενιαία πληρωμή σκοπεύουν εκεί να εφαρμόσουν ένα σύστημα ίδιας πληρωμής που ήδη συμπεριλαμβάνει μια ανακατανομή και δεν θέλουν περαιτέρω ανακατανομή και έχουν μια επιπλέον αντίρρηση επί της αρχής. Έχουν μια προσέγγιση αν θέλετε ελευθέρου εμπορίου και η έννοια δηλαδή των συνδεδεμένων επιδοτήσεων δεν τους βρίσκει σύμφωνους. Γι' αυτό δεν ε, εφαρμόζεται. Αυτός είναι ένας λόγος. Και από ό,τι καταλαβαίνω εγώ επιτρέπεται σε μια χώρα σαν τη Φιλανδία που πάντα η, έλεγε πως ε, δεν ε, ήταν σωστή ευρωπαϊκή πολιτική για τις συνθήκες Φιλανδίας να ε, σε επέτρεπε να προσαρμόσει την πολιτική αυτή. Οπότε υπάρχει μια κάποια ευελιξία χωρίς να επιβάλλει σε όλους ε, να εισαχθεί ένας τέτοιο μηχανισμός. Η κυρία Μαγκίνε τώρα μίλησε για τη δικαιοσύνη. Έχει δίκιο. Δεν νομίζω. Ε, Τέλο πάντων, το μόνο σχόλιο μπορώ να κάνω είναι πως ε, η δράση της γαλλικής κυβέρνησης, το να μειώσει δηλαδή την ενιαία πληρωμή και να εφαρμόσει το άρθρο 63, μάλλον έχουν ε, επιφέρει περισσότερη δικαιοσύνη, όπως θα το βλέπει τουλάχιστον ένας οικονομολόγος, στο γαλλικό σύστημα, από δράσεις που είχαν αποτελέσει στο παρελθόν αντικείμενο κριτικής σε σχέση με τους μεγάλους αγρότες. Οπότε νομίζω το συγκεκριμένο ζήτημα το αντιμετώπισε το γαλλικό κράτος με το άρθρο 63 και 68. Εάν υπάρχουν άλλες χώρες ε, οι οποίες θεωρούν πως υπάρχει ζήτημα δικαιοσύνης, ε, τότε αυτοί είναι μηχανισμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διορθώσουν την κατάσταση. Αλλά βεβαίω η εφαρμογή του συστήματος αυτού κατά αποκοπήν ε, πληρωμής ε, νομίζω πως θα αντιμετωπίσει πολλές από τις αντιρρήσεις περί δικαιοσύνης. Τώρα δεν είμαι σίγουρος για το τα σχόλια αρκετών βουλευτών για την πολιτική. Ήταν σχόλια, δεν, δεν μπορούσα να απαντήσω εγώ σε αυτά. Εάν έχετε όμως κάποιες ερωτήσεις ε, για να εξετάσουμε, έχουμε ακόμα τρεις εβδομάδες ε, πριν ολοκληρώσουμε τη μελέτη μας, οπότε αν έχετε συγκεκριμένα σχόλια ή πράγματα τα οποία δεν περιέχονται στην έκθεση, Ε, που δεν σας τα είπαμε εμείς και θα μπορούσαμε να σας τα πούμε ευχαρίστως να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πιτ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για αυτή την ε, δυνατότητα που μας δώσατε να παρέμβουμε σε αυτήν την τόσο σημαντική μελέτη. Τώρα, πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο, τον κύριο Ντάσιαν Σόλος. Του δίνω, τον καλωσορίζω λοιπόν ευθύς αμέσως. Μετά την ακρόαση του Ιανουαρίου είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο και θα συζητήσουμε στο πιο σημαντικό ντοσχέ αυτής της ε, θητείας που είναι το τι θα γίνει για την ΚΑΠ μετά το 2013. Θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται άμεσες απαντήσεις για να, για βγει από την κρίση. Εμείς ε, θελήσαμε να καταθέσουμε μία προφορική ερώτηση με ψήφισμα για τα μελλοντικά μέσα διαχείρισης της αγοράς που θα συζητηθεί στο Στρασβούργο στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα. Είμαι σίγουρος ότι ο Επίτροπος Τσόλος και την επόμενη εβδομάδα θα μας δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα με το μέλλον της ΚΑΠ και θα συζητήσουμε την έκθεση του κυρίου Τζόρζ Λάιον που όπως πολλές φορές επαναλάβαμε είναι ε, μια εξαιρετική βάση για τις εργασίες μας το λόγο ευθύς αμέσως ο Επίτροπος, μετά ο εισηγητής και μετά οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Στη συνέχεια η συζήτηση θα είναι απόλυτα ανοιχτή. Λοιπόν, Ντάτσαν έχεις το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Πάολο. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής ε, που σας συναντώ εδώ. Πριν από Μερικούς μήνες είχα έρθει, αλλά ήμουν καθισμένος εκεί κάτω. Τώρα, όπως είδατε, ε, ψήλωσα, ανέβηκα. Θυμάμαι τις πρώτες ανταλλαγές που είχαμε και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε κατά τον ίδιο τρόπο. Εγώ εκμεταλλεύομαι αυτήν την ε, πρώτη μου τοποθέτηση ε, μετά, πρώτη τοποθέτηση μετά το διορισμό μου για να σας μιλήσω για το μέλλον της ε, ΚΑΠ και ευχαριστώ τον Πάολο Δικάστρο για την πρόσκληση όπως και τον George Λάιον για τις ε, ε, εργασίες του σχετικά με την έκθεση για το μέλλον της ΠΑΚ. Γνωρίζετε ότι θα πρέπει να γράψουμε μία νέα σελίδα για την ΚΑΠ μετά το 2013 και αυτήν τη σελίδα θα τη γράψουμε μαζί. Εγγράφεται απόλυτα στο πλαίσιο της στρατηγικής που πρότεινε η Κομισιόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εν ώψη του 2020. Ε, συγγνώμη. Θεωρώ ότι η Γεωργία μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην ευφύη ανάπτυξη, στην αηφόρο ανάπτυξη και η στρατηγική του 2020 προβλέπει μία ευθυγράμμιση της ΚΑΠ με τους οικονομικούς μας στόχους. Σας το είπα και πριν ότι για μένα είναι η πρώτη μου προτεραιότητα να ξαναγράψω αυτές τις σελίδες για το 2020. Ο παππούς μου ήταν χωρικός, αγρότης, στην ε, βορειοανατολική Ρουμανία. Και η σοφία του με συνόδεψε σε όλες τις φάσεις της ζωής μου και έμαθα πολλά πράγματα και για τη γεωργία και για τη ζωή. Και έλεγε μια παλιά παροιμία που φαντάζομαι ότι και σε, άλλες, ε, σε άλλους ευρωπαϊκούς ε, πολιτισμούς ότι πολλές φορές το δέντρο κρύβει το δάσος. Και πολλές φορές ε, θυμάμαι εγώ αυτή την παροιμία, αυτό το απόφθεγμα όταν σκέφτομαι την ΚΑΠ. Ο καθένας τελικά κοιτάει το δέντρο του και λίγοι κοιτάνε το δάσος. Έτσι ξεκίνησε και η συζήτηση για την ΚΑΠ. Μια συζήτηση πολύ ζωντανή, αυτό είναι καλό πράγμα, διότι σημαίνει ότι η Γεωργία ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά προχωράμε πολλές φορές πολύ πιο γρήγορα από όσο χρειάζεται. Ξεψηρίζοντας τις λεπτομέρειες και αγνοώντας το δάσος. Εγώ ξέρω έχοντας μεγαλώσει κοντά σε ένα Γιώργο τι σημαίνουν αυτές οι λεπτομέρειες για πολλούς ότι τους αρέσουν. Αλλά θυμίζω ότι το δέντρο πολλές φορές κρύβει το δάσος. Πρέπει πάντα να κρατάμε μία απόσταση, να έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας για να μπορούμε να διαμορφώνουμε τις απόψεις μας και να σχεδιάζουμε. Γιατί πρέπει να δούμε σε τι χρειάζεται αυτό το δάσος που είναι η ΚΑΠ. Συμβολικά μιλάω. Αυτό να ρωτιέστε κι εσείς και εγώ το ίδιο να ρωτιέμαι. Και ρωτώ και όλους τους πολίτες σχετικά. Επιστήμονες, καταναλωτές, φορολογούμενους, εμπόρους, γεωργούς, βιομηχάνους, Πιστεύω ότι και οι Ευρωπαίοι πρέπει να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα και πρέπει να το σκεφτούν σοβαρά πριν μπουν σε λεπτομέρειες. Η Ευρώπη είναι υπεύθυνη για την ε, αυτάρκεια των πολιτών της. Και η Λισαβόνα επαναλαμβάνει αυτήν την ανάθεση ευθύνης. Και αυτό ήταν και ο στόχος της Τρέζα το 1958 όταν ε, τέθηκαν τα θεμέλια της ΚΑΠ. Τότε είχαμε πολλά δέντρα αλλά δεν είχαμε γεωργικές μηχανές. Ε, και ονειρευόταν η Ευρώπη ε, να ξεπεράσει την λογική του επισητισμού και του συσιτίου. Ήθελε λοιπόν τροφιμική ασφάλεια και αυτή η ανάγκη παραμένει. Τα τελευταία γεγονότα των τελευταίων ετών μας το θυμίζουν. Πρέπει να είμαστε περήφανοι λοιπόν για ό,τι έγινε. Αλλά θα πρέπει να έχουμε και τη δύναμη και τη σοφία να προχωρήσουμε μέσα σε μια Ευρώπη 27 κρατών που είναι ένα πιόνι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παγκοσμιοποιημένου κόσμου. Οι αποφάσεις μας θα έχουν επιπτώσεις, σοβαρές επιπτώσεις ε, προς τους πολίτες μας στην καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ατόμων και στην Ευρώπη αλλά και αλλού. Οι αποφάσεις μας δεσμεύουν και το μέλλον ενός ευρωπαϊκού σχεδίου. Οι πολίτες είναι πολλές φορές σκεπτικιστές για αυτά τα, γύρω από αυτά τα σχέδια και το χαμηλό ποσοστό της συμμετοχής στις τελευταίες ευρωεκλογές κάτι τέτοιο αποδεικνύει. Πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να γίνει ορατή και να αποκτήσει υπόσταση. Οι πολίτες εκφράζουν ανησυχίες, ερωτηματικά και προσδοκίες που πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας. Πρέπει λοιπόν να συμμετέχουν οι πολίτες όταν εμείς παίρνουμε αποφάσεις. Οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν τι γίνεται εδώ, στα κέντρα συζητήσεων και αποφάσεων. Η ΚΑΠ είναι μια πολιτική κλειδί στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση και ολοκλήρωση και η ΚΑΠ είναι και πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική σήμερα. Σίγουρα υπάρχουν κριτικές, ε, γίνονται κριτικές, υπάρχουν ατέλειες. Αλλά υπάρχουν και προσδοκίες και πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας όχι για να αποδυναμώσουμε ή να καταργήσουμε την ΚΑΠ. Το λέω, το βροντοφωνάζω αυτό. Πρέπει να την καταστήσουμε πιο ισχυρή για τους Ευρωπαίους γεωργούς σήμερα, να είναι ένα μέσο δηλαδή αυτή η πολιτική για το μέλλον, όχι ένα εργαλείο του παρελθόντος. Εγώ είμαι υπέρ της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ εν του 2013 και θεωρώ ότι υπάρχουν τρεις λόγοι τουλάχιστον για να γίνει κάτι τέτοιο. Πρώτο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μια συνεκτική και συλλογική απάντηση μέσα από τη στρατηγική του 2020 και για να απαντήσει δηλαδή στην οικονομική και δημοσιονομική κρίση, για να αντιμετωπίσει τις κλιματικές αλλαγές και να ανακάμψει την οικονομική ανάπτυξη ενισχύοντας και τον ανταγωνισμό. Η ΚΑΠ συμβάλλει σε όλα αυτά, διότι αποτελεί κλειδί της δύναμης μυκής της υπαίθρου και αποτελεί κινητήρα για τη ζωτικότητα της υπαίθρου μας. Η ΚΑΠ συνδέεται με την Ευρώπη 2020 και είναι αναπόσπαστο κομμάτι για μία υφόρο ανάπτυξη. Δεν μπορούμε εμείς να μιλάμε για λογική χρήση των φυσικών πόρων χωρίς να έχουμε κατά νου τη γεωργία. Η ΚΑΠ είναι απαραίτητη και για την απασχόληση επιτρέπει στην Ήπεθρο να αναπτύξει πλήρως το δυναμικό της. Και ξέρουμε ότι η γεωργική απασχόληση βρίσκεται στη βάση σε αυτές τις περιοχές και άμα δεν υπάρχει γεωργία δεν υπάρχει και δουλειά. Η ΚΑΠ είναι απαραίτητη και για την πράσινη ανάπτυξη. Και όταν ασκείται ισορροπημένα δίνει απάντηση στις κλιματικές αλλαγές. Η ίδια γεωργία αποτελεί πηγή ανανεώσιμης ενέργειας. Εμπνέει για την ευφύ ανάπτυξη. Και πρέπει εμείς να φανταστούμε και στο, για το μέλλον πώς θα γίνει αυτή η ευφύης ανάπτυξη δηλαδή να παράγουμε παραπάνω με λιγότερους πόρους, φυσικούς πόρους. Να μειώσουμε τις ε, εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακος, τις εκπομπές που δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η εφής ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει παραμερίζοντας ε, τη Γεωργία και δεν μπορεί και η Γεωργία να αναπτυχθεί χωρίς αυτή την αντίληψη. Σήμερα είμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση 27 κρατών μελών και κάθε κράτος μέλος είναι διαφοροποιημένο και ως προς τον πολιτισμό και ως προς τη γεωργία. Είναι ένα πλούτος για όλους μας και ιδίως για τους γεωργούς. Πρέπει να ενισχύσουμε τη σχέση μεταξύ γεωργών και καταναλωτών, μεταξύ της παραγωγής της εντόπιας και των αγορών σε τοπικό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να μιλάμε πια για ένα μοναδικό ευρωπαϊκό υπόδειγμα στη γεωργία. Δεν είναι ομοιογενής πια η γεωργία μας, αλλά είναι πολύμορφος και πολυσχηδής. Δεν έχουμε μία λοιπόν γεωργία μονάχα, αλλά πολλές γεωργίες στην Ευρώπη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας λοιπόν αυτή την πολυμορφία και τον πλούτο που εκπροσωπεί. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα διατηρηθεί και θα χρησιμοποιηθεί για το καλό όλης της κοινωνίας μας. Αλλά η διατήρηση αυτής της πολυμορφίας δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επανέλθουμε σε εθνικού χαρακτήρα πολιτικές σε βάρος μιας κοινοτικής πολιτικής στον τομέα της γεωργίας γιατί αν δεν μπορούμε να δούμε το σύνολο είναι πολύ πιο δύσκολο, είναι σχεδόν αδύνατο να διαχειριστούμε τα συστατικά του τμήματο. Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια συνολική αντιμετώπιση και μόνο μια ευρωπαϊκή πολιτική στο τομέα της γεωργίας μπορεί να διατηρήσει την πολυμορφία της γεωργίας. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη να καταγράψουμε αυτή την πολυμορφία και να προσαρμόσουμε την κοινή μας πολιτική σε αυτή την πολυμορφία για να υπάρχει καλύτερη διαχείριση τις ποικιλία στο γεωργικό τομέα. Τρίτον, χρειάζονται και προσαρμογέ γιατί πρέπει να προετοιμάσουμε το μέλλον. Θα πρέπει να επιτρέψουμε στη γεωργία να ανταποκριθεί στι προκλήσει τη κοινωνία σήμερα. Τροφιμική ασφάλεια, προστασία των εδαφών, των φυσικών πόρων, οικονομική ανάπτυξη στους ε, αγροτικούς τομείς, κλιματική αλλαγή. Οι πολίτες και οι φορολογούμενοι θα κατανοήσουμε τον τρόπο αυτό ότι η κοινή αγροτική πολιτική είναι προς το συμφέρον τους. Δεν πρέπει να θεωρηθείτε ότι είναι ένας τομέας πολιτικής που αφορά μόνο τους γεωργούς, γιατί όλη η κοινωνία ευνοείται από την κοινή αγροτική πολιτική με καλύτερα τρόφιμα και καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια έλλειψη επαφών της κοινής αγροτικής πολιτικής με τους Ευρωπαίους πολίτες. Πριν από μερικές εβδομάδες μια έρευνα του Ευρωμαρόμετρου έδειξε ότι πάνω από 90% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρούν ότι είναι σημαντική η γεωργία για το μέλλον. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Πάνω από 90% των Ευρωπαίων περιμένουν από τη γεωργία να τους δώσει ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα και υψηλής ποιότητας. Να προστατεύσει επίσης η γεωργία το τοπίο, το περιβάλλον, να είναι πηγή ανάπτυξης οικονομίας. Εδώ υπάρχει απόλυτη σύμπνοια των Ευρωπαίων πολιτών. Αλλά δείχνει αυτό, η, μάλλον η έρευνα, ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν ξέρουν πολύ καλά τι είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Μόνο ένας από τους σε κάθε τρεις Ευρωπαίους ξέρει κάτι για το τι είναι η κοινή αγροτική πολιτική, ποιο είναι το περιεχόμενό της ποια είναι η εφαρμογή της. Είναι εύγλωτα λοιπόν αυτά τα στοιχεία, πολύ πιο εύγλωτα από ό,τι θα μπορούσα να σας πω εγώ. Ο λίγων κατ' ο λίγων η ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική έχει γίνει υπόθεση των επαϊών των μονάχα, των εμπειρογνωμόνων. Θα πρέπει να ανατρέψουμε αυτή την τάση και να φέρουμε και πάλι σε επαφή με τον πληθυσμό την κοινή αγροτική πολιτική. Πρωτού προχωρήσουμε σε μια μεταρρύθμιση, θα πρέπει να θέσουμε σωστά τα ερωτήματα και να τα συζητήσουμε. Θα πρέπει να εμπλέξουμε του πολίτε και την κοινότητα των πολιτών, να του δώσουμε την ευκαιρία και το χώρο και τον χρόνο να εκφράσουν την άποψή τους, ώστε συνέχεια να λάβουν υπόψη τις απόψεις που θα συλλέξουμε στις μελλοντικέ πρωτοβουλίες μας με έναν τρόπο που θα είναι συνεκτικός. Και γι' αυτό τονίζω την ανάγκη να υπάρξει μια δημόσια συζήτηση σε σχέση με το ρόλο της γεωργίας στην κοινωνία της Ευρώπης, σε σχέση με το ρόλο και τη θέση της γεωργίας και σήμερα και αύριο. Και για το ποιοι είναι οι στόχοι που πρέπει να εξυπηρετηθούν από την κοινή αγροτική πολιτική. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτή η άσκηση και δεν είναι μια περίτη άσκηση. Προτού λοιπόν συζητήσουμε για τα εργαλεία, για τον προπολογισμό, για τα προγράμματα και όλα αυτά. Προφανώ υπάρχουν χώροι όπου πρέπει να ληφθούν κάποιε αποφάσει. Θα πρέπει όμω να έχουμε το χρόνο να ακούσουμε την άποψη των απλών ανθρώπων προτού περάσουμε σε μια επίσημη διαδικασία λήψη απόφαση. Αν δεν επενδύσουμε το χρόνο για να υπάρξει αυτό ο προβληματισμό και η ευρύτερη συζήτηση, ο κίνδυνο θα είναι να μιλάμε για τα μέσα μια πολιτική που ακόμα δεν θα έχουμε καθορίσει ή που θα έχουμε καθορίσει μονάχα μεταξύ των εμπειρογνώμων. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξει μια ευρεία και ελεύθερη συζήτηση με όλου του συμπολίτε μα. <clears throat> γιατί θέλουμε μια ευρωπαϊκή γεωργία, γιατί μια κοινή αγροτική πολιτική. Και κατά τη διάρκεια αυτή τη συζήτηση μπορούμε να συλλέξουμε τι απόψει και τι θέσει όλων των εμπλεκομένων. Τι ιδέε αυτών που θέλουν να συμμετάσχουν είτε με μονομένα σε άτομα, είτε μέσω ενώσεων, παραγωγών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, δεξαμενών σκέψη ή οποιοδήποτε άλλο φορέα. Εγώ περιμένω λοιπόν να έχουμε τι απόψει των γεωργών κυρίως, των επαγγελματικών του ενώσεων, αλλά επίση και των φορέων προστασία του περιβάλλοντο, των ενώσεων αυτών, των καταναλωτών, των ενώσεων που υποστηρίζουν την ευζοία των ζώων όλων αυτών που ασχολούνται για τον τομέα της ε, ασφάλειας των τροφίμων, της βιώσιμης ανάπτυξης ή της αγροτικής ανάπτυξης. Τα θέματα σε σχέση με το μέλλον που θα πρέπει να απαντήσουμε είναι πολλαπλά. Υπάρχουν πολλές πτυχές οι οποίες θα πρέπει να τύχουν ανάλυσης. Για μένα <clears throat> αρθρώνεται η συζήτηση αυτή γύρω από τέσσερα στρατηγικά ερωτήματα. Πρώτον, γιατί θέλουμε μια κοινή αγροτική πολιτική. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλά επιχειρήματα, θα πρέπει να τα διατυπώσουμε και να είναι σαφή και ιδίως να τα ακούσουμε και από μη εμπειρογνώμονες. Δεύτερον, ποιοι είναι οι κοινωνικοί στόχοι για την, ε, οι στόχοι της κοινωνίας μας για τη γεωργία με όλη την πολυμορφία της. Τρίτον, γιατί θα πρέπει να υπάρξει μια μεταρρύθμιση τη τωρινή κοινή αγροτική πολιτική και πώς μπορεί να γίνει με έναν τρόπο ο οποίος ανταποκρίνεται στι προσδοκίε τη κοινωνία μα. Τέταρτον, ποια είναι τα εργαλεία τα οποία θα απαιτηθούν για τη μελλοντική μεταρρύθμιση κοινή αγροτική πολιτική για κάθε ένα από αυτά τα ερωτήματα προκύπτουν και άλλα ερωτήματα τα οποία θέλω να τα επισκοπήσω τώρα. Πρώτον, με ποια εργαλεία μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της επιστηστικής ασφάλειας η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί στο μέλλον θα έχουμε μια επιτάχυνση και μια διαφοροποίηση της παγκόσμιας ζήτησης για τρόφιμα. Έχουμε χώρες οι οποίες αναδύονται και χώρες οι οποίες θα πληγούν από την κλιματική αλλαγή. Δεύτερον, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι ο καταναλωτής έχει προϊόντα υψηλής ποιότητα ασφαλή σε προσβάσιμες τιμές. Πώς θα το εξασφαλίσουμε αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συγχρόνω θα καλύψουμε τις ανάγκες των τοπικών περιφερειακών αγορών και του αγροτροφημικού τομέα. Πώς θα εξασφαλίσουμε την πράσινη και αηφόρο οικονομική ανάπτυξη στους χώρου τη υπαίθρου. Αυτέ οι περιοχέ μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο και σε οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο απασχόληση και προστασία του περιβάλλοντο. Πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα εργαλεία που είναι προσαρμοσμένα στι περιοχέ αυτέ, είτε είναι ε, περιαστικέ περιοχέ, είτε όχι, οι οποίε έχουν μεγάλο παραγωγικό δυναμικό και χωρίς ένα ισχυρό αγροτικό τομέα θα απειληθεί η οικονομία του. Τέλο, ποιο θα είναι το κληροδότημά μα στις μελλοντικέ γενναίε σε σχέση του περιβάλλοντος, ποιότητος αέρος, εδαφών και ύδατος. Οι γεωργοί που είναι λιγότερο από 5% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαχειρίζονται και αξιοποιούν περίπου το 80% του ευρωπαϊκού εδάφους. Πώς λοιπόν θα διαχειριστούμε καλύτερα τους φυσικούς πόρους, ενώ παράγουμε αγροτικά προϊόντα. Πώς θα διατηρήσουμε και τη βιοποικιλότητα του ευρωπαϊκού χώρου. Περαιτέρω, η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια ένα θεωρητικό ερώτημα. Η κοινωνία περιμένει και από τον αγροτικό τομέα να υπάρξουν λύσει για την κλιματική αλλαγή και έχει δείξει ήδη η Γεωργία ότι μπορεί να δώσει απαραίτητε απαντήσει για την μείωση ιδίω τη εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Υπήρξε μία μείωση κατά 20% στην εκπομπή των αερίων αυτό μεταξύ του 1990 και του 2007, ενώ στην σύνολη οικονομία, σε όλου του οικονομικού τομεί, η μείωση ήταν μονάχα 8%. Ακόμα μπορούμε να πράξουμε πολλά. Αλλά εκεί θα πρέπει να έχουμε μια πιο στενή σύνδεση μεταξύ έρευνα και γεωργία για να βρούμε του καλύτερου τρόπου να το κάνουμε αυτό. Επίση, ποιο μέλλον θα πρέπει να έχει η Ευρώπη στι διεθνεί αγορέ. Ποια είναι τα ισχυρά μα σημεία, πώ θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα τα σημεία που έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Πώ μπορούμε να έχουμε ποιοτικέ προδιαγραφέ που να είναι όσο και πιο δυνατόν ανοιχτέ σε τρίτε χώρε. Σε σχετικά, σχετικά με το θέμα αυτό, σα δίνω μοναχά ένα παράδειγμα. Το θέμα τη ευζοία των ζώων. Θα πρέπει λοιπόν από αυτές τις προκλήσεις να προκύψει η... ο σκελετός μιας πολιτικής η οποία θα υποστηρίξει την αηφόρο γεωργία και το περιβάλλον. Και πρέπει επίσης να θέσουμε και περαιτέρω ερωτήματα. Πώς θα δημιουργήσουμε εργαλεία τα οποία θα είναι πιο ορατά για τον ε, καταναλωτή, ώστε να καταλαβαίνει τη σχέση μεταξύ αγροτικής υποστήριξης και την ε, λειτουργία των αγορών και των ε, διανομέων των αγροτικών προϊόντων. Με ποια εργαλεία θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα ενός ελάχιστου εισοδήματος για τους γεωργούς πώς θα πρέπει να είναι οι επιδοτήσεις προς τους γεωργούς και πώς πρέπει να γίνονται με ένα ισοδικαίο τρόπο. Πώς θα απαντήσουμε στην μεγάλη διακύμανση που έχουν πολλές φορές οι αγορές βασικών προϊόντων. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι μια οικονομική κρίση δεν μπορεί να οδηγήσει στον όλεθρο ένα ολόκληρο οικονομικό τομέα. Πώς θα μπορέσουμε να έχουμε ισορροπημένες σχέσεις μεταξύ των διαφόρων οικονομικών συντελεστών στον αγροτοτροφημικό τομέα. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι ο καταναλωτής καταβάλει ένα λογικό τίμημα για τα αγροτικά προϊόντα και επίση έχουν ένα δίκαιο και αξιοπρεπέ εισόδημα και οι Γεωργοί πώ θα εξασφαλίσουμε ότι η πολυμορφία τη γεωργία στην Ευρώπη θα διατηρηθεί και στο μέλλον και πώ θα μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη τα ιδιαίτερα προβλήματα τα οποία προκύπτουν για να αντιμετωπίσουμε την ανταγωνιστικότητα αυτή τη γεωργία και τι είδους ανταγωνιστικότητα θα προωθήσουμε σε αυτέ τι περιπτώσει. Ποιε είναι οι απαντήσει που έχουν να κάνουν με την περαιτέρω ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα, δηλαδή τη ανάπτυξη του αγροτροφινικού τομέα σε δεύτερο επίπεδο, πώ θα μπορέσουμε να δώσουμε δυναμική στην οικονομία μα μέσω τη πράσινη ανάπτυξη. Πώ θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και του ανθρώπου και φυσικού πόρου τη περιοχή τη Υπέθρου και πώ θα μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε την απερίμωση ορισμένων περιοχών. Και τέλο, ποια είναι η αγροτική πολιτική και η Ευρώπη τη γεωργία που θέλουμε εμεί να αφήσουμε στα παιδιά μα στο μέλλον. Ξέρω λοιπόν ότι όλα αυτά είναι πάρα πολλά ερωτήματα. Έχω θέσει πάρα πολλά ερωτήματα και σήμερα. Έχουμε κάποιους μήνες στη διάθεσή μας για να δώσουμε μια απάντηση προτού φτάσουμε στην υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων. Και η δημόσια συζήτηση που σας ζητώ να συμμετάσχετε σε αυτή ξεκινάει και θα κρατήσει, προτείνω, μέχρι τον Ιούνιο του 2010. Αυτός ο χρονικός ορίζοντας θα μας επιτρέψει, πιστεύω, να διευκρινίσουμε αυτά που περιμένει η Ευρώπη σε σχέση με τη Γεωργία. Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι παρόν σε όλα τα κράτη-μέλη, σε διάφορες εκδηλώσεις που θα οργανωθούν, όπως και οι συναδελφοί μου. Θα είμαι παρόν επίσης και στην Επιτροπή των Περιφερειών και στην ΟΚΕ για να παρουσιάσω τις ιδέες σε σχέση με αυτή τη δημόσια συζήτηση. Από σήμερα υπάρχει μια ιστοσελίδα μέσα στη σελίδα της Κομισιόν, στον χώρο της Κομισιόν για αυτούς που θέλουν να κάνουν προτάσεις και θα υπάρξει και μια σύνθεση όλων αυτών των προτάσεων από έναν εξάρτητο οργανισμό και στη συνέχεια τον Ιούνιο, 19 και 20 Ιουνίου προβλέπεται να διοργανωθεί μια μεγάλη συνδιάσκεψη εδώ στις Βρυξέλλες που είσαστε φυσικά καλεσμένοι για να αντιληφθούν τα συμπεράσματα από αυτή τη μεγάλη δημόσια συζήτηση ώστε να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη στην συνέχεια της συζήτησης. Ελπίζω λοιπόν ότι μέχρι το τέλος του έτους θα μπορεί η Κομισιόν να έχει υποβάλει μια ανακοίνωση για τους στόχους της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής και θα μπορέσει να υπάρξει και μια συνεκτική συζήτηση των προτάσεων αυτών. Γιατί πεπισμένο είμαι ότι θα βρούμε νέες καινοτόμε και ισχυρέ ιδέες οι οποίες μπορούν να προέρχονται από τους πολίτες, από τους εμπλεκόμενους στον αγροτικό τομέα, από αυτούς που θα είναι οι κύριοι αποδέκτες αυτήν την πολιτική. Βασίζομαι λοιπόν στην υποστήριξή σας για αυτή τη διαδικασία γιατί εσείς έχετε την ευκαιρία να έχετε μια πιο άμεση επαφή με τη βάση, με τους απλούς πολίτες και ελπίζω θα υπάρξουν και συνεισφορές από τη δική σας πλευρά αλλά και από αυτούς που συναντάτε σε εκλογικές σας περιφέρειες. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σας και ελπίζω ότι δεν σας έκανα να βαρεθείτε με όλα αυτά που σας είπα. Μου φάνηκε ότι ήταν σημαντικό να χρησιμοποιήσω αυτή την παρουσία με ενώπιόν σας για να σας παρουσιάσω αυτή τη δημόσια συζήτηση και εξάλλου είναι απαραίτητο να έχουμε και μια συζήτηση στη συνέχεια για το εξαιρετικό έργο του George Lyon. Και είμαι έτοιμο φυσικά να απαντήσω τα ερωτήματά σα και να συζητήσω για οποιαδήποτε αυτά τα θέματα. Σα ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ αγαπητέ Επίτροπε. Ξεκινάμε τη συζήτηση. Θα είναι μια συζήτηση πολύ ουσιαστική, βλέποντας δηλαδή και τον αριθμό των ε, εγγεγραμμένων ομιλητών. Γι' αυτό παρακαλώ να είστε σύντομοι για να εκμεταλλευτείτε και το χρόνο ομιλία. Ο Τζόρτζ έχει αμέσως το λόγο γιατί είναι εισηγητής και μετά θα μιλήσουν οι συντονιστές των ομάδων. Τζόρτζ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον Επίτροπο που ήρθε σήμερα στην Επιτροπή μας και παρουσίασε την ε, δημοσία συζήτηση η οποία θα ξεκινήσει και βεβαίω για τα σημαντικά ερωτήματα που έθεσε που θα μας απασχολήσουν τους επόμενους μήνες. Βεβαίω η συζήτηση αυτή δεν θα μπορούσε να έρθει σε καταλληλότερη στιγμή γιατί ελπίζουμε μέχρι τον Ιούλιο όταν θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια την έκθεση ε, Πρωτοβουλία ε, την οποία έχουμε ήδη μπροστά μα μπορεί νομίζω να συνεισφέρει στην διαβούλευσή σα και να δώσει κάποιε απαντήσει. Θα είμαι σύντομο. Θα τονίσω κάποια πράγματα που είναι στην έκθεσή μου γιατί ξέρω πως και οι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Μου έκανε εντύπωση κάτι το οποίο είπε στην αρχή ο Επίτροπος που είπε πως είναι ένα σημαντικό εργαλείο για το μέλλον η κοινή γεωρική πολιτική και όχι του παρελθόντος. Πραγματικά η κυνηγιογική πολιτική μόλις μεταρρυθμιστεί πρέπει να είναι η λύση και οι απαντήσεις για το μέλλον και όχι να αναπολύει το παρελθόν. Και νομίζω πως στο εγγραφό μου ε, προτείνω ένα όραμα με το οποίο μπορούν οι αγρότες να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του 21ου αιώνα και στις απαιτήσεις κοινωνίας. Κατόπιν ο Επίτροπος στις παρατηρήσεις του ανέφερε κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Η μεγαλύτερη νομίζω είναι ο διπλασιασμός της ζήτησης για παραγωγή τροφίμων μέχρι το 2050. Μια τεράστια πρόκληση γιατί αυτή τη φορά δεν γίνεται να ανοίξει αν θέλετε η κάνουλα όπως το παρελθόν. Τον σπαταλάμε ενέργεια και λιπάσματα και ζανιοκτώνα δεν θα είναι κάτι που θα μπορούμε να κάνουμε λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ε, οι ευρωπαϊκές γέες πρέπει να συνεισφέρουν σε αυτή τη λύση και να παράγουν βέβαια περισσότερο τρόφιμα. Υπάρχει ζήτημα διαθεσιμότητας του νερού και η μεγαλύτερη πρόκληση είναι βεβαίως η ακριβή ενέργεια και ίσως και η έλλειψη ενέργειας. Και αυτό βεβαίως ε, σημαίνει πως θα είναι δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά την παραγωγή τροφίμων σε σχέση με τα προηγούμενα 60 χρόνια, όταν και πάλι διπλασιάστηκε η παραγωγή τροφίμων. Αυτή νομίζω είναι η μεγάλη πρόκληση. Η μεγάλη αύξηση της ζήτησης, η διατροφική ασφάλεια θα εξακολουθεί να παίζει μεγάλο ρόλο μετά το 2015, αλλά πρέπει να δούμε και την κλιματική αλλαγή, την πράσινη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, τις νέες αυτές προκλήσεις της ε, στρατηγικής ε, του 2020. Και πρέπει να πούμε πως η γεωργία είναι απάντηση, είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Στο δέγγραφο μου αναφέρω τις βασικότερες ε, προτεραιότητες για μια δικαιότερη αηφόρο και πιο πράσινη γεωργία, κοινή γεωργική πολιτική. Και νομίζω πως η δικαιοσύνη εδώ πέρα είναι σημαντικό γιατί πρέπει να υπάρχει και αηφορία. Δεν μπορούμε, όπως είπα, να συνεχίσουμε να βάζουμε πόρους ε, στη γη και να αναμένουμε απλά ε, παραγωγή. Πρέπει να υπάρχει αηφορία στο μέλλον και η κοινή γεωργική πολιτική είναι το μέσο για να επιτευχθεί αυτό. Όπως είπα και η δικαιοσύνη είναι βασικός παράγων της μεταρρύθμισης κοινή γεωργικής πολιτικής. Όταν λέω δικαιοσύνη εδώ πέρα μιλάω για δίκαιο εμπόριο ε, για τους αγρότες έναντι καλά επιδοτούμενων εμπορικών εταίρων. Θα πρέπει να παίζει επίσης όρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους εταίρους μας και αυτό είναι βασικό τμήμα του τι θα γίνει μετά το 2013 και αυτό ισχύει και για τις εισαγωγέ που έρχονται. Πρέπει να υπάρχει και εκεί πέρα δικαιοσύνη για τους Ευρωπαίους αγρότες. Αυτό σημαίνει βέβαια και δικαιοσύνη έναντι όλων των χωρών που έχουν μεγάλη καλλιεργήσιμη γη που είναι οριακή. Πρέπει να υπάρχει παραγωγή τροφίμων και γεωργική δραστηριότητα σε όλη την Ευρώπη. Επίσης πρέπει να υπάρχει μια δίκαιη πληρωμή των αγροτών, επίσης δικαιοσύνη στη διατροφική αλυσίδα, θα μπορούν δηλαδή οι παραγωγοί να μπορούν να ζήσουν καλύτερα, μεγαλύτερη διαφάνεια στη διατροφική αλυσίδα, να δουν πού γίνονται οι καταχρήσεις, να κατονομάσουμε και να ντροπιάσουμε όσους δεν ανταγωνίζονται σωστά και να υπάρχει μια ελάχιστη ασφάλεια στο σύστημα, δηλαδή σε καιρούς κρίση να μπορούμε να διασφαλίσουμε πως υπάρχει σταθερότητα και όχι τόση αναταραχή όσο είδαμε πρόσφατα. Επίσης πιστεύω πως μέρος αυτής της δικαιοσύνης είναι να δούμε τις ανισχύες των νέων κρατών μελών για την κατανομή των κονδυλίων. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό το ερώτημα και το αναφέρω στην έκθεσή μου. Υπάρχουν εκεί πέρα κάποιες προτάσεις. Ένα σημαντικό ζήτημα εδώ πέρα είναι να διασφαλίσουμε και να δούμε πώς θα υπάρχει δικαιοσύνη των παλαιών κρατών σε σχέση με τα νέα και πώς θα το επιτύχουμε αυτό. Επίσης η αηφορία πρέπει να είναι στην καρδιά της κοινής γεωργικής πολιτικής. Προσπάθησα να την εντάξω στις ε, προτάσεις ε, που κάνω στα πέντε αυτά βασικά κομμάτια. Όπως είπατε και ο ίδιος η Γεωργία ήδη έχει επιδείξει την δυνατότητα να μειώσει τις εκπομπές. Πρέπει λοιπόν ε, να διασφαλίσουμε πως μπορεί η Γεωργία να κάνει περισσότερα και με καλύτερο τρόπο. Η εφορία πρέπει να είναι στην καρδιά της παραγωγής τροφίμων και η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να διασφαλίσει πως θα το προωθήσουμε αυτό στο μέλλον. Αυτό σημαίνει και αποτελεσματικότητα της παραγωγής, γιατί δεν είναι θέμα μόνο περιβαλλοντικό, αλλά και οικονομικό, θέμα οικονομικής αηφορίας. Και οπωσδήποτε στο μέτωπο της κλιματικής αλλαγής έχουμε ένα διπλό όφελος. Έχουμε και περιβαλλοντική αηφορία και οικονομική αηφορία μέσω κάποιων μέτρων που προτείνω για την κλιματική αλλαγή και βεβαίως η προστασία του περιβάλλοντος. Μια πρασινότερη κυνήγική πολιτική πρέπει να δούμε πως τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα θα καλύπτουν πολύ περισσότερη έκταση από ό,τι αυτή τη στιγμή για να βοηθήσουμε και τη βιοπικιλότητα. Επίσης έχουμε εδώ πέρα και την πράσινη ανάπτυξη. Να Δοθώσουμε κίνητρα έτσι ώστε οι αγρότες να μπορέσουν να γίνουν παραγωγή πράσινης ενέργειας μέσω βιομάζας, βιοαερίου, απέ μικρής κλίμακας. Πρέπει λοιπόν και η κυνηγυρική πολιτική να δώσει εκεί πέρα όθηση, γι' αυτό ζητάμε πιο δίκαιη, πιο πράσινη και πιο αηφόρο κυνηγυρική πολιτική. Έχω ορίσει λοιπόν τα πέντε βασικά σημεία που μπορούν να δώσουν αυτά τα αποτελέσματα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Τα βασικά νομίζω στοιχεία που πρέπει να υποστηρίξουμε για το μέλλον είναι πρώτον άμεσες πληρωμές που θα διασφαλίζουν διατροφική ασφάλεια και δίκαιο εμπόριο. Δεύτερον, εθνικές ε, συμπληρωματικές ε, στρεματικές ε, πληρωμές που θα δώσουν κίνητρο για, την κλιματική αλλαγή, για τη βελτίωση αποτελεσματικότητας και την περιβαλλοντική και οικονομική αηφορία ταυτοχρόνως, θεμελιώδες κατά την άποψή μου, η γεωργία σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι μειονεκτικές περιοχές ε, ε, παραμένουν Ω βασικό στοιχείο τη κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2013, βιοπικιλότητα και προστασία του περιβάλλοντο τέταρτο πυλώνα, για να διασφαλίσουμε πω τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα θα καλύπτουν σημαντικό περισσότερη έκταση από ό,τι στο παρελθόν για να βελτιωθεί η βιοπικιλότητα και η προστασία του περιβάλλοντος και πέμπτο κομμάτι η πράσινη ανάπτυξη, η δυνατότητα που μας δίνει η γενιά της πράσινης ενέργειας για να μπορέσουν οι αγρότες να βρουν και άλλες πηγές εισοδήματο με τις νέες αυτές τεχνολογίες. Τα πέντε αυτά λοιπόν στοιχεία θα πρέπει βεβαίως να στηρίζονται σε ένα ελάχιστο δίκτυο ασφαλείας, να υπάρχει μια ελάχιστη στήριξη όταν δεν υπάρχει δυνατότητα απορρόφηση από την αγορά, να έχουμε κάποια μέσα ε, άμεσης αντίδρασης και επίσης ζητώ να δούμε την πολιτική ανταγωνισμού. Μήπως δηλαδή θα μπορέσουν οι ενώ των αγροτών να διαπραγματευτούν καλύτερα την τιμή των προϊόντων τους. Να δούμε επίσης ε, την ε, αγορά των futures των συμβολέων μελλοντικής ε, εκπλήρωσης για να χρησιμοποιηθούν ίσως στο μέλλον. Αυτά για μένα είναι τα πέντε βασικά στοιχεία με το δίκτυο ασφαλείας όπως σας είπα. Ελπίζω πως τις συζητήσεις θα έχουμε διακομματική στήριξη για κάποιες από τις ιδέες που ανέφερα. Η έκκλησή μου είναι να μην μπούμε στις λεπτομέρειες σε αυτό εδώ το έγγραφο, γιατί εδώ πέρα αναφέρουμε τις αρχές, τις προτεραιότητες, όχι τις λεπτομέρειες του πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Γιατί αν καταλήξουμε με χίλιες τροπολογίες για το κάθε ζήτημα, οι Κομισιόν θα διαλέξουν όποιες ε, θέλουν και θα πούνε «Α, εμείς ε, ό,τι θέλατε κάναμε». Αυτά και ελπίζω οι συνάδελφοι να δουν το θέμα επικοδομητικά για να καταλήξουμε σε μια θέση η οποία θα είναι συνεκτική, αξιόπιστη και θα διασφαλίσει το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Grazie Molto bene. Πολύ καλά, Τζόρτζ, ευχαριστώ. τέλα παρόλα. Ο Άλμπερτ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Επίτροπο Τσιόλος και τον κύριο Λάιον. Εγώ, συντονιστής της ομάδος μου, θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα σημεία. Εμείς αναρωτιόμαστε κύριε Επίτροπε αν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Παλιά παντούσε η Επιτροπή τα ερωτήματά μας. Τώρα εσείς μας θέσατε πάρα πολλά ερωτήματα και δεν έχουμε στην πραγματικότητα το χρόνο να τα απαντήσουμε. Ίσως λοιπόν θα μπορούσα να ζητήσω να απαντήσετε και μερικά ερωτήματα εσείς ο ίδιος. Για την έκθεση George Lyon να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτά που παρουσίασε και μπορώ να συμφωνήσω με πολλά από αυτά τα οποία λέει ο εισηγητή. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιε παρατηρήσει οι οποίε εν καιρό θα πρέπει να συζητηθούν στην Επιτροπή μα. Για μένα είναι ορθό, κύριε Επίτροπε, και εσείς να υποστηρίξετε τη διατήρηση ενός πρώτου πυλώνα και στο μέλλον της Γεωργίας, νομίζω ότι αυτό το αναφέρει και ο Τζορτς Λάιον, ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια προσαρμογή για τα νεα κρατημέλη και θα πρέπει να γίνει με σταδιακό τρόπο αυτή η προσαρμογή. Αυτό βέβαια μπορεί να αποτελέσει και σημείο συζήτηση στο μέλλον. Εγώ θεωρώ πολύ θετική την έκθεση του κυρίου Λάιον. Αντιμετωπίζει πολλά από τα θέματα τα οποία εδώ θα μπορέσουμε στην Επιτροπή μας να τα συζητήσουμε πιο ενδελεχώς. Θέλω να υποστηρίξω απόλυτα τον εισηγητή επίσης στην ε, αίτησή του να διατηρηθεί και μετά και επέκεινα το 2013 η χρηματοδότηση της Γεωργίας γιατί μια Ευρώπη των 27 ή αύριο των 28 κρατών μελών δεν μπορεί να λειτουργήσει με λιγότερα κονδύλια για την Γεωργία. Υποστηρίζω περαιτέρω τον εισηγητή όταν λέει ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία επιστροφή στις ε, ε, συνδεδεμένες ε, επιδοτήσεις και θα πρέπει να διατηρήσουμε μονάχα σε μερικές εξαιρετικές περιπτώσεις μια ελάχιστη μορφή σύνδεσης. Όπως λέει ο εισηγητής θα πρέπει να υπάρξουν νέες παράμετροι για την απόδοση άμεσων επιδοτήσεων και όχι μονάχα η αρρώσιμη επιφάνεια. Μπορούμε να συζητήσουμε περαιτέρω υποδείγματα. Επίσης για να διατηρήσουμε την ε, ανταγωνιστικότητα της γεωργίας θα πρέπει να μην εξασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα μόνο Θα πρέπει να δούμε ποια ακριβώς θα πρέπει να είναι η μελλοντική μας αγροτική πολιτική. Κατανοώ κύριε Επίτροπε ότι εσείς δεν θέλετε να διατηρήσετε το τωρινό επίπεδο στον πρώτο πυλώνα, αλλά συγχρόνως Ακόμα και αν αυτό είναι σημαντικό στις διαπραγματεύσεις των διαπραγματεύσεων για τον ΠΟΕ, το να έχουμε δηλαδή μια ανταγωνιστικότητα στον τομέα αυτό, θα πρέπει εξάλλου να εξασφαλίσουμε και μια ανταγωνιστικότητα επί τη βάση υψηλότερων προδιαγραφών στη Γεωργία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμεί μπορούμε να το υποστηρίξουμε και ενώπιον των πολιτών μας. Το να έχει η Ευρωπαϊκή Γεωργία ένα υψηλό επίπεδο προτίμων. Νομίζω ότι υπάρχει μια ευρεία συνένεση για κάτι τέτοιο. Συμφωνούμε όλοι ότι ένας από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωση είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε για μισό δισεκατομμύριο ανθρώπων προσβάσιμα και υψηλής ποιότητα γεωργικά προϊόντα. Και αν κατάλαβα καλά αυτά που λέτε κύριε Επίτροπε, σωστά, είπατε ότι 80% της ε, επιφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στην διαχείριση των γεωργών. Και αυτό είναι κάτι το αξιοσημείο ότι 5% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να διαχειριστούν τα 80% της έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την έκθεση του George Lyon έχω κάποιες αμφιβολίες για την ιεράρχηση των διαφόρων στοιχείων, για την απαρίθμηση των στοιχείων αυτών Νομίζω ότι αυτά τα οποία ανέφερε στο τέλος της εκθεσής του ίσως θα πρέπει να θεθούν σε υψηλότερο επίπεδο. Στην αρχή της έκθεσής του δηλαδή, σε ό,τι αφορά το μέλλον της αγιορικής πολιτικής μετά το 2013. Κύριε Επίτροπε, θα πρέπει, πιστεύω, να δώσουμε προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή ευθύνη, την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 27 κράτη-μέλη και να κρατήσουμε σε δευτερεύον επίπεδο τα εθνικά συμφέροντα. Λοιπόν, θα πρέπει με γνώμονα τα ευρωπαϊκά και όχι τα εθνικά συμφέροντα να μπορέσουμε να εξεύρουμε μια καλή συμβαστική λύση η οποία θα εξασφαλίσει το μέλλον και των γεωργών επέκεινα του 2013. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι γεωργοί και όχι μόνο οι επιχειρήσει θα έχουν καλές προοπτικές στην Ευρώπη μετά από το 2013 και η δική μου πολιτική ομάδα θέλει να εμπλακεί πλήρω σε, αυτή την, σε αυτό το εγχείρημα που αναφέρατε για την δημόσια διαβούλευση και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και εμείς τη συνεισφορά μας στην έκθεση George Lyon. Ευχαριστώ Άλμπερτ, ο Λουίς ε, Κάπουλα Σάντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να απευθυνθώ καταρχήν στον κύριο Επίτροπο, να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του και να υπογραμμίσω ότι οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες υποστηρίζουν ιδιαίτερα το ύφος με το οποίο εκτελεί το έργο του, διατηρώντας μια πολιτική ανεξαρτησία που είναι αξιοσημείωτη και επίση ένα ανοιχτό πνεύμα για να ακούσει την άποψη όχι μόνο των πολιτικών αλλά και των Γεωργό, και του γεωργού και τι οργανώσει του. Ο κύριο Επίτροπο μα πρότεινε μια μεθοδολογία και μα έθεσε και μια πλειάδα ερωτήματων. Εγώ πρέπει να πω ότι συμφωνούμε με τη μέθοδο και θέλουμε να συμμετάσχουμε με δέσμευση και ενθουσιασμό στο εγχείρημα αυτό διαβούλευση. Θέλω να σα υπενθυμίσω όμω ότι πρέπει και εμείς να δώσουμε μια απάντηση στις προσδοκίες και τις ανησυχίες αυτών που μας έχουν στείλει εδώ των εκλογέων μας και θα πρέπει λοιπόν και ενώπιον αυτών των πολιτών να είμαστε σε θέση να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσε ο κύριος Επίτροπος για την έκθεση του κυρίου Λάιον και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λάιον για την εργασία του και για τον τρόπο με τον οποίο έχει λειτουργήσει μαζί με τους συναδέλφους, ιδίως τους συντονιστές και θα ήθελα εδώ απλώς να αναφερθώ στις θετικές πτυχές της έκθεσής του για την πρώτη αυτή μορφή της έκθεσής του και τις πτυχές που θεωρώ λιγότερο ευτυχής. Νομίζω ότι είναι πολύ εύληπτη και ευανάγνωστη η έκθεση του κυρίου Λάιον και εγώ Χαίρομαι για την πράσινη απόχρωση που διατρέχει αυτή την έκθεση και είναι μια πολύ καλή συνεισφορά σε αυτήν την ε, προβληματική. Ζητά να υπάρχει οπωσδήποτε απαράγραπτα μια ευρωπαϊκή ε, γεωργία. Δέχεται να υπάρχει αυτή η στρεματική ενίσχυση και φυσικά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ρόλος των γεωργών που παρέχουν ένα δημόσιο αγαθό δέχεται ότι μπορεί να υπάρχει μια επιφυλακτική μετάβαση από το υπάρχον σύστημα σε ένα νέο σύστημα και θεωρεί θετικά όλα αυτά τα οποία έχει διαγράψει η Κομισιόν σε επίπεδο προτεραιοτήτων και θεωρώ ότι η πρότασή του για ένα πέμπτο άξονα, αυτό που αναφέρει ως πράσινη ανάπτυξη, είναι πάρα πολύ θετική. Ο εισηγητής διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος των αγρο αγροτοπεριβαλλοντικών ε, μέτρων για την Ευρωπαϊκή Γεωργία, υποστηρίζει τις μειονεκτικές περιοχές, δίνει πρόσθετες επιδοτήσεις για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι προσπάθειες για την αναχέτηση της κλιματικής αλλαγής και η εκθεσή του είναι εξάλλου πάρα πολύ ανοιχτή για να μπορέσουν να υπάρξουν και επιπλέον συνεισφορές. Από την άλλη πλευρά όμως, και αναφέρομαι στα λιγότερα θετικά θέματα, Νομίζω ότι χρειάζεται μια προβλημα... ένα περισσότερο προβληματισμός για ορισμένα θέματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην, στην έκθεση. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για τις ε, ενισχύσεις επί τη βάση της ε, καλλιεργούμενη επιφάνεια υποστηρίζει τις λεγόμενες οικολογικές πτυχές μονάχα. Επίση, δεν αναφέρεται καθόλου στην ε, προϋπόθεση μιας ελάχιστης Δραστηριότητα των γεωργών. Αυτό έρχεται σε αντίφαση με αυτά τα οποία διαπραγματεύτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΠΟΕ και ίσως η Κομισιόν θα μπορούσε να μας πει αν πράγματι υπάρχει ασυμβατότητα αυτής της πρότασης με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΠΟΕ. Και επίσης ο εισηγητής μιλάει για ισοδίκαια μεταχείριση. Δεν εξηγεί όμως ποια είναι η μηχανισμοί που θα προτείνει για να προωθήσει αυτή την δικαιοσύνη. Και συγχρόνως εισάγει κάτι το οποίο ανησυχεί, λέει ενισχύσεις ανά εκτάριο αλλά θα πρέπει να τροποποιούνται, να διαμορφώνονται επί τη βάση ενός συντελεστή αγοραστικής δύναμης των γεωργών. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι μεγαλύτερη η, ε, η επιδότηση στους γεωργούς της χώρας που έχουν μικρότερη ε, αγοραστική δύναμη, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αυτός είναι και ο στόχος του εισηγητή. Επίσης νομίζω ότι βασίζεται σε υπερβολικό βαθμό στην συγχρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο ζητάνε είναι κάτι που ξεπερνάει το τωρινό υπόδειγμα της κοινή γεωργικής πολιτικής και αυτό είναι ασύμβατο με την τωρινή κατάσταση οικονομικού οικονομικό επίπεδο πολλών κρατών μελών που δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν μια τέτοια συγχρηματοδότηση. Αυτό θα σημαίνει ότι θα υπάρξει μια ανισότητα μεταξύ των πιο πλουσίων και πιο ασθενών κρατών μελών και επίσης προτείνει ήδη, και αυτό είναι υπερβολικό αυτή τη στιγμή, ένα προϋπολογισμό για την κοινή αγροτική πολιτική που να είναι στο επίπεδο του 2013. Όταν λοιπόν βάζει κανείς την μπάρα τόσο ψηλά, σημαίνει ότι θα δεχτεί σε συμβαστικό επίπεδο μια χρηματοδότηση κάτω από αυτήν που θα είναι του 2013. Εμείς το λέμε από τώρα, δεν μπορούμε να δεχτούμε χρηματοδότηση υποδέστερη αυτή του προπολογισμού του 2013. Επομένω, δεν είναι καλή η διαπραγματευτική θέση του εισηγητή. Λέει επίση ο εισηγητή πάρα πολλά για την απλοποίηση σε όλη την ε, έκθεσή του για το υπόδειγμα ε, το οποίο προτείνει. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν είναι αποτελεσματικές προτάσεις, θα πρέπει εμείς με τις τροπολογίες μας να προτείνουμε ουσιαστική απλοποίηση. Επίσης δεν βλέπω κάποια αναφορά στη συνέχιση των κοινωνικο-οικονομικών επιδοτήσεων για την ε, δασοκομεία, παραγωγή για την προστασία της ε, πολυμορφίας στις οικονομικές δραστηριότητες, μίς όπου εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί η έκθεσή του. Και εξάλλου, Το υπόδειγμα του κύριου Λάιον μου φαίνεται ότι είναι μια συνέχεια του παρελθόντος, ότι δεν είναι αρκετά καινοτόμο. Υπήρχαν βέβαια οι θετικέ αυτές πτυχές που ανέφερα προηγουμένως ότι τονίζει την πιο πράσινη ανάπτυξη, αλλά δεν αποκλίνει αρχικά αρκετά από το τωρινό υπόδειγμα. Εμείς ως σοσιαλιστές θέλουμε περισσότερα πράγματα και στην απλοποίηση του υποδείγματο και στην απλοποίηση και στην ε, καινοτομία. Θέλω, εν πάση περιπτώσει, να, εξάρω τον ρόλο του κυρίου Λάιον και τη θαυμάσια εργασία του, που είναι μια πολύ καλή βάση εργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λουίς. Ο Μάρτιν Όσλιν, συνόμιλος των Πρασίνων. Ε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Είναι η πρώτη μεγάλη συζήτηση που κάνουμε. Ευχαριστώ και τον Τζόρτς για την έκθεση. Δεν ξέρω, φαίνεται πως εδώ πέρα κάνουμε ερωτήσεις, αλλά νομίζω πως ε, θα πρέπει να κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις για να λάβουμε τις σωστές απαντήσεις. Εγώ θεωρώ πως ένα μου προξένησε εντύπωση, κανένας δεν χρησιμοποίησε πλέον την έκφραση ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο. Ποια είναι η διαφορά μας από τους άλλους, ποια είναι τα πλεονεκτήματά μας και που πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε αυτά. περιγράψαν πολύ θετικά την κατάσταση και έχουμε αγνοήσει προβλήματα που υπάρχουν όντως. Αν ρωτούσαμε τους αγρότες θα έλεγαν πως ε, δεν, δεν είναι δυνατή η κατάσταση. Το είπε ο Τζόρτζ. Ε, τα γεωργικά εισοδήματα παραμένουν ε, χαμηλά σε σχέση με αυτά τα οποία χρειάζονται. Οπότε αυτό είναι μέρος του προβλήματος και αν δεν δώσουμε λύση δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε άλλο με αυτό το ζήτημα, να τα παρατήσουν οι αγρότες. Κάτι το οποίο φαίνεται ήδη και υπάρχει σε πολλές περιοχές. Ε, ολόκληρα χωριά ερημώνουν. Επίσης, ε, ένα ερώτημα σε σχέση με την έκθεση Μιλάμε για το ζήτημα της κατανομής της δίκαιης κατανομής των μέσων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο ζήτημα κατανομής μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και εντός της γεωργίας. Δηλαδή, προς στιγμή, ε, αυτή τη στιγμή επωφελούνται οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις παρά οι μικρότερες, ε, παρά το ότι βεβαίως εκεί πέρα βρίσκονται οι περισσότερες θέσεις εργασίας. Πρέπει να το πούμε αυτό πρέπει το σύστημα να παραμείνει ως έχει. Είναι βάση για τις ε, μελλοντικέ ε, ε, εξελίξεις και αν επαρκεί μόνο η πολλαπλή συμμόρφωση για τις πληρωμές και συνέχεια λέμε ότι πρέπει να έχουμε μια πιο ανταγωνιστική γεωργία και πολιτική αλλά ο ανταγωνισμός και οι στόχοι της ανάπτυξης πρέπει να οριστούν ξανά. Το βλέπουμε στον τομέα του γάλακτος το μισό, των, το 50% των επιχειρήσεων χάθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια και αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση θα χάσουμε και άλλες. Με κρατικές ενισχύσεις μιλάμε, συνέχεια. Οπότε ποιος είναι ο στόχος αυτής της πολιτικής, ποιος είναι ο στόχος αν στο δεύτερο πυλώνα, παραδείγματο χάρη ασχολούμαστε μόνο με την ανταγωνιστικότητα και στη γεωργία Βλέπουμε πως ε, σβήνουν, χάνονται πολλές επιχειρήσεις και μαζί τους θέσεις εργασία. Πρέπει λοιπόν να ορίσουμε ξανά τους στόχους γεωργικής πολιτικής ως στόχους που θα δέχεται και η κοινωνία. Αναφέρθηκε η κλιματική αλλαγή. Όχι αρκετά. Η γεωργία είναι τμήμα της λύσης αλλά και του προβλήματος. Δεν πρέπει να το κρύβουμε τι κάνουμε. Εμείς μετατοπίζουμε τις εκπομπές μας στον τρίτο κόσμο, από όπου λαμβάνουμε τις ζωοτροφές. Κόβουμε τα τροπικά δάση στη, Βραζιλία για να καλλιεργηθούν προϊόντα που έρχονται εδώ πέρα. Αυτό δεν μπορεί να το χρεώνεται μόνο η Βραζιλία. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Να δούμε το κρίσιμο ερώτημα που είπε ο Τζόρτζ στην αρχή, το θέμα της παγκόσμιας διατροφής. Το δικό μας το μοντέλο είναι ε, αυτό το οποίο μπορεί να συνεισφέρει. Ε, δεν ξέρω, εγώ αναρωτιέμαι. Γιατί νομίζω πως έτσι ξεχνάμε το ότι με τη δική μας γεωργία, με αυτόν τον τρόπο γεωργίας, δεν μπορούμε να διαθρέψουμε 90, ε, με 9 δισεκατομμύρια ανθρώπους, γιατί θα καταντήσουν το φαγητό να είναι είδος πολυτελείας. Επίσης, δίνουμε το σωστό μήνυμα προς την ε, νέα γεωργική πολιτική. Εδώ πέρα πρέπει να πω πως ε, εξεπλάγει λίγο για το ότι τα πρώτα μηνύματα της Κομισιόν στον τομέα της γεωργίας ήταν η, η έκρηση ε, γενετικά τροποποιημένης πατάτας. δεν είναι και πολύ θετικό μήνυμα για την πρόοδο της γεωργίας να μιλάμε για γενετική τεχνολογία πάλι. Πρέπει να το πούμε Εάν θέλουμε ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο, πρέπει να υπάρχει διάκριση από τα γεωργικά μοντέλα άλλων χωρών. Πρέπει να λάβουμε σοβαρά την συνύπαρξη, να μιλάμε για οικολογική γεωργία. Χρειαζόμαστε γεωργία με δικαιώματα των αγροτών και μια γεωργία που θα είναι οικολογική. Πιο οικολογική. Ο Τζόρτζ ε, χρησιμοποιεί τη λέξη, μιλάει για μια πιο πράσινη ε, γεωργία, αλλά δεν υπάρχει ουσία εδώ πέρα. Επίσης είπατε πως χρειαζόμαστε μια ευρύτατη συζήτηση. Αυτή πράγματι χρειάζεται, όχι μόνο να συζητάμε μεταξύ αγροτών, να συζητήσει όλη η κοινωνία πράγματι. Και εδώ πέρα βέβαιως συμπεριλαμβάνονται και οι καταναλωτές. Οπότε πρέπει και αυτοί να συμπεριληφθούν και βεβαίως πάντα με ένα ευρωπαϊκό μέτρο. για τη γεωργία στον Ευρώπη. Στην ποικιλία της αλλά και στην ενότητα και εμείς θέλουμε να συνεισφέρουμε σε αυτό και στις ε, συζητήσεις ε, που θα έχουμε για να έχουμε μία κοινή γεωρική πολιτική που θα την αποδέχονται όλοι. Ε, ευχαριστώ Μάρτιν. Για τους συντηρητικούς, σε έχει το λόγο. <coughs> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήταν πολύ θετικό αυτό που άκουσα κύριε Επίτροπε. Δεν είναι η πρώτη φορά που σας ακούμε να τοποθετήσετε. Και η... το όραμά σας για την ΚΑΠΑ είναι αποδεκτό στην Επιτροπή μας. Αλλά τα πάντα εξαρτώνται από το τι συμβαίνει έξω από αυτή την αίθουσα. Φτάνει λοιπόν μόνη τη η πολιτική βούληση της Κομισιόν για να μορφοποιήσει την ΚΑΠ. Πολύ μ' άρεσε εμένα αυτή η μεταφορά που κάνατε, να μην βλέπουμε μόνο το δέντρο, να κοιτάμε το δάσος. Σήμερα χρειαζόμαστε μια διαφορετική πολιτική. Δεν πρέπει απλώς να περιορίσουμε το δάσος, πρέπει να το ξαναφυτέψουμε. πρέπει να το ξαναφυτέψουμε, είναι πιο μεγάλη σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε μια πολιτική πιο διευρυμένη. Ο κύριος Λάιον και άλλοι ομιλητές ανέφεραν το τι μας περιμένει στο μέλλον. Χρειαζόμαστε περισσότερα τρόφιμα Χρειαζόμαστε λοιπόν μια πιο ισχυρή ΚΑΠ. Κύριε Επίτροπε, υπάρχει ένα πρόβλημα εξομοίωσης των πληρωμών. Και πρέπει ήδη σήμερα να υποδείξουμε πώς θα έχει η κατάσταση μετά το 2013. Λοιπόν, πώς μπορούμε εμείς να κάνουμε τη σύγκριση λέγοντας ότι θα προηγούνται τα νέα κράτη-μέλη και τα παλιά κράτη-μέλη ακολουθούν. Ποιο είναι το συγκριτικό μέτρο για όλα αυτά. Χρειάζονται λοιπόν διαφορετικές τοποθετήσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Εμείς σήμερα Μιλήσαμε για τη συνθήκη της Λισαβόνας και όλοι ήταν πανευτυχείς. Όταν όμως όλοι μιλά, ε, φτάνουμε στη συζήτηση του προϋπολογισμού, τόσο περισσότερο εθνικιστές γινόμαστε. Πρέπει να αλλάξει λοιπόν αυτή η τοποθέτηση. Πρέπει να είμαστε ευρωπαϊστές και για τη συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά και για τον προϋπολογισμό. Η ΚΑΠ χρειάζεται λεφτά. Χωρίς λεφτά δεν κάνουμε τίποτα. Ο κύριος Λεγέρικ. Α, δεν είναι. Είναι, είναι. Κύριε Επίτροπε, κύριε Λάιον, σας ευχαριστώ για τις τοποθετήσεις σας. Όπως είπατε κύριε Επίτροπε υπάρχει μια γενική φιλοσοφία η οποία διέπει τις ιδέες σας αλλά υπάρχει όμως και μια βάση αρκετά ανησυχητική ένα φόντο ανησυχητικό. Πιστεύω ότι υποτιμάτε το γεγονός ότι σήμερα η ύπεθρος βιώνει ένα δράμα. Το μέσο γεωργικό εισόδημα είναι χαμηλότατο, έχετε πολλούς γεωργούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι έχουν ξεπεράσει πλέον το κατόφλι της παινίας και έχουμε, μια, έχουμε χρέωση και υπερχρέωση των γεωργικών επιχειρήσεων. Αυτό δεν το είπατε πουθενά και χρειάζονται κατεπήγοντα μέτρα, διότι αλλιώς ε, τίνουμε προς μια πραγματική κοινωνική καταστροφή και η οποία θα είναι βέβαια και μια χωροταξική καταστροφή. Συμμερίζομαι τη γενική φιλοσοφία που διέπει τις θέσεις σας κύριε Επίτροπε και αυτές του κυρίου Λάιον όπως και μέρος των αναλύσεων που κάνετε. Αλλά υπάρχει ένα πρώτο ζήτημα και πρέπει να αναρωτηθούμε υπάρχει πάντοτε μία πραγματική ΚΑΠ ή ενότητα των τιμών, η δημοσιονομική ιδρυτική ισχυρότητα. Αυτές οι, οι, οι ιδρυτικές αρχές υφίστανται. Εγώ δεν το πιστεύω. Και ποιες είναι οι επιπτώσεις του γεγονότος ότι δεν υφίστανται πλέον αυτές οι αρχές. Έχουμε δραματικές επιπτώσεις από την απουσία τους. Σας τα ανέφερα προηγουμένων. μείωση των τιμών, ε, μείωση των εισοδημάτων και μεταφορά του κόστους ε, είτε προς το φορολογικό σύστημα είτε προς ε, τον καταναλωτή. Και ποιος κερδίζει από όλα αυτά οι πολυεθνικές γενικώ και οι ευρωπαϊκές πολυεθνικές ειδικότερα. Έχουμε λοιπόν γενική υποβάθμιση των συνθήκων ζωής των μικρομεσαίων αγροτών. Φοβούμε λοιπόν ότι για μια ακόμη φορά αναφέρεται ελάχιστα αυτό το θέμα και εσείς και στην έκθεση του κυρίου Λάιον. Δηλαδή ουσιαστικά προσαρμόζουμε τη γεωργία σε ένα διεθνές σύστημα, αυτό που μας επιβάλλει ΠΟΕ. Έχουμε λοιπόν, λέω, μία προσαρμογή της ΚΑΠ στους κανόνες που μας επιβάλλει η Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου με όλες τις επιπτώσεις που θα επιφέρει κάτι τέτοιο για τη μικρομεσαία γεωργία. Υπάρχει ένα μόνιμο επιχείρημα που έρχεται και, και επανέρχεται, δηλαδή ότι πρέπει να, να ταΐσουμε τον κοσμάκι. Αλλά το να αναπτύξουμε εμείς μία υπηρωτική πολιτική λέγοντας ότι πρέπει να ταΐσουμε τον κοσμάκι, μα τότε πραγματικά εμείς εδώ θα υποσκάψουμε την τροφιμική ανεξαρτησία και της υπήρου μας αλλά και των άλλων υπήρων. Όταν, όταν αναλύουμε τα πράγματα, τι βλέπουμε, βλέπουμε ότι συνεχώς συμπιέζονται οι τιμές. Δηλαδή άμα η πρεμούρα μας είναι, μία, είναι ο ανταγωνισμός σε μία ανοιχτή αγορά, τότε τι θα γίνει, θα μας ξεφύγει η κατάσταση και θα, και θα έχουμε αυτά τα δράματα τα οποία γνωρίζουμε σήμερα, τα οποία είναι και κοινωνικά δράματα και περιβαλλοντικά. Ε, ε, ε, δράματα. Εμείς ε, Εμείς δεν έχουμε ένα δικό μας σχέδιο για την πρωτεΐνη, συνεχίζουμε να εισάγουμε σόγια ή μανιόκα. Δεν ασκούμε μια πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος με αυτές τις καλλιέργειες και έχουμε ένα τεράστιο, τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος που δεν είναι καν μετρήσιμο για την κοινωνία. Πολύ σωστά όλα αυτά τα ερωτήματα που θέτετε κύριε Επίτροπε. Θα συμμετέχουμε εμείς στη συζήτηση. Θα το κάνουμε ως κοινωνία των πολιτών και όπως και οι άλλες ομάδες θα το κάνουνε. Και αυτό για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην προσέγγιση των στόχων που εσείς ο ίδιος θέσατε. Ευχαριστώ κύριε Λεράκ. Το λόγο στον Επίτροπο για να δώσει μία πρώτη απάντηση στους συντονιστές και μετά θα συνεχίσουμε με τις 17 ε, επόμενες ε, τοποθετήσεις και μετά θα ολοκληρώσει ο Επίτροπος. Αγαπητέ Ντάσαν, έχεις το λόγο. Εγώ θέλω να τονίσω μετά από αυτές τις υποθέσεις που άκουσα ότι εντάξει έχουμε το μέλλον αλλά έχουμε και το παρόν και οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν στους γεωργούς αλλά για τις απαντήσεις που χρειάζονται άμεσα δεν μπορούμε να περιμένουμε το 2014 πρέπει να απαντήσουμε κάτι και τώρα. να έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα επανέλθω βέβαια και στο τέλος της συζήτησης για την έκθεση αυτή. Είναι μια έκθεση την οποία εσείς θα την αναπτύξετε περαιτέρω, θα την εξευγενήσετε. Ο George Lyon έχει κάνει εξαιρετική εργασία και ίσως θα πρέπει να κλείσει αυτό στη συζήτηση για το θέμα αυτό. Μπορώ να σας δώσω μερικές ε, ιδέες, αλλά καταρχήν θέλω να απαντήσω στην ανησυχία σας σε σχέση με το παρόν πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να κοιτάμε το μέλλον και να ξεχνάμε το παρόν. Να κοιτάμε τα δέντρα και να μην βλέπουμε το δάσος λοιπόν, να χάσουμε τη γενική εικόνα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν μια ισορροπία σε ό,τι αφορά τα μέτρα αυτά. Για τα άμεσα μέτρα τώρα, ξέρετε, εγώ αναφέρθηκα ήδη στο γαλακτοκομικό τομέα Όπου από τη μία πλευρά αντιμετωπίσαμε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο επηρέασε ιδιαίτερα το εισόδημα των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων, αλλά και μας οδήγησε στη συνειδητοποίηση ότι χρειάζεται να υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί οι οποίοι τώρα ελείπουν ώστε να μπορέσει να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στο γαλακτοκομικό τομέα. Το είπα και ενώπιον του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας πρόσφατα. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε το 2013 για να προτείνουμε λύσεις για τα θέματα αυτά. Θα χρησιμοποιήσω όλες τις δυνατότητες που έχω στη διάθεσή μου αυτή τη στιγμή και η ομάδα υψηλού επίπεδου για τα γαλακτοκομικά θα παρουσιάσει τα πόρισματά της Οσονούπο. Θα υπάρξει μια συζήτηση λοιπόν στη συνέχεια στο Συμβούλιο Υπουργό και θα μπορούσαμε να έχουμε και μια συζήτηση μαζί σας και στη συνέχεια αυτών ζήτησα από τις υπηρεσίες μου να καταρτήσουν ένα πακέτο μέτρων μέχρι το τέλος του ενεστώτος έτους για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα διορθωτικά μέτρα αυτά το ταχύτερα δυνατόν. Να εφαρμόσουμε λοιπόν τα πορίσματα τα οποία είναι εφαρμόσιμα τη ομάδα υψηλού επίπεδου για το γάλα και για όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την σύναψη συμφωνιών, με την κατανομή του εισοδήματος και των εσόδων σε όλο αυτό το τομέα. Αν υπάρξει η δυνατότητα μιας απάντησης σε ρυθμιστικό επίπεδο θα το πράξουμε και σας διαβεβαιώνω ότι ακόμα κι αν εγώ θέλω να επικεντρωθώ στα θέματα του μέλλοντος, παρακολουθώ από κοντά και την εξέλιξη των αγορών στην περίπτωση που υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να κάνουμε κάποιες ε, τροποποίησεις. Για να επανέλθω τώρα εν συντομία στον πρώτο αυτό γύρο παρεμβάσεων από τους συντονιστές. Νομίζω ότι το κατανοείτε ότι δεν είναι η στιγμή που εγώ θα μπορέσω να σας δώσω επακριβείς και λεπτομεριακές απαντήσεις σε σχέση με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία εγείρονται από την έκθεση George Lyon. Το είπα και στην εισαγωγή μου, θα το πω και τώρα. Είναι μια ευχάριστη έκπληξη για μένα η ποιότητα των παρεμβάσεων που έχουν γίνει, Όλα ουσιαστικά τα θέματα τα οποία πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας έχουν αντιμετωπιστεί, όλα τα θέματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν στην προετοιμασία της μεταρρύθμισης. Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες, υπάρχουν τομείς όπου χρειάζεται περισσότερη εξέλιξη, αλλά όπως είπε και ο Ζόρζ, το πιο σημαντικό είναι να μην προχωρήσουμε βεβαιασμένα για να δούμε τι είδους μηχανισμούς θα έχουμε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σωστά το χρόνο μας για να κατανοήσουμε πρώτα ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι μας και τι προστοκούμε από τη μεταρρύθμιση που θα επιφέρουμε στην κοινή αγροτική πολιτική. Για να πάρω το παράδειγμα των αμέσων πληρωμών. Σίγουρα τίθεται το θέμα μιας ισοδίκαιας κατανομής των επιδοτήσεων. πόσα θα πάρουμε από τον ένα χώρο και πόσα θα δώσουμε στον άλλο. Με ποια ταχύτητα θα γίνει η μετάβαση από το ένα σύστημα πληρωμών στο άλλο. Αλλά εξάλλου είναι και πιο σημαντικό να δούμε ποιος είναι ο στόχος αυτών των αμέσων επιδοτήσεων. Είναι σημαντικό για μας για να μπορέσουμε να λάβουμε μία απόφαση, αλλά είναι σημαντικό να είναι σαφές και για τον καταναλωτή. Γιατί δίνουμε άμεσες επιδοτήσεις στους γεωργούς. Γιατί στο μέλλον δεν θα είναι αντισταθμιστικές πληρωμές όπως ήταν στο παρελθόν, με ιστορικές αναφορές. Δεν θα υπάρχει αυτός ο αντισταθμιστικός και μόνον χαρακτήρας, θα είναι αναμένοντας και αμείβοντας μία δραστηριότητα από του γεωργού, την οποία παρέχουν ήδη μέσω τη αγροτική του δραστηριότητα. Επομένω, το ερώτημα είναι τι θέλουμε να επιτύχουμε με τι άμεσε αυτέ επιδοτήσει από κάθε μορφή γεωργία, από κάθε είδο γεωργών, από κάθε αγροτικό τομέα. <clears throat> Και με αυτή την εκκίνηση, αυτό το σημείο αφετηρίες μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς με τον απλούστερο δυνατό μηχανισμό. Συμφωνώ λοιπόν ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας μια τροποποίηση του συστήματος που θα το απλοποιήσει. Θα πρέπει όμως συγχρόνως να δούμε τι ακριβώς επιζητούμε με τις άμεσες επιδοτήσεις για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει και κάποιο αντιστάθμισμα στον εισόδημα των γεωργών, αλλά επίσης να παροτρύνουμε τους γεωργούς για την παροχή ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών και να αντιμετωπίσουμε και τη μειονεκτική μορφή ορισμένων περιοχών, να διατηρήσουμε θέσει απασχόληση. Νομίζω λοιπόν ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποιο είναι το ειδικό βάρο όλων αυτών των επιμέρου ε, στοιχείων για να μπορέσουμε να καθορίσουμε ποιο θα είναι και το επίπεδο των αμέσων επιδοτήσεων. Κατά τα άλλα τώρα, για την απλοποίηση. Και στην περίπτωση αυτή πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν, αλλά κυρίως με γνώμονα μια ισορροπία μεταξύ της διοικητικής απροποίησης, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία των πληρωμών και των οικονομικών υποστηρίξεων να γίνεται μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, αλλά όχι μόνο σε διοικητικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο αναγνωσιμότητας, δηλαδή να είναι σαφείς αυτοί οι μηχανισμοί και εύκολοι να τους κατανοήσει κανείς. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στο θέμα της συνεκτικότητος μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα ή αν θέλετε μεταξύ των επιδοτήσεων που έχουμε για, ε, για το εισόδημα και την αμοιβή για την παροχή ενός δημοσίου αγαθού. Επομένως μεταξύ υποστήριξης, το εισόδημα και της, του εξυγχρονισμού της γεωργικής δραστηριότητα και επίσης θα λάβουμε, πρέπει να λάβουμε υπόψη της μη οικονομικού χαρακτήρα δραστηριότητα στον τομέα της, στον χώρο των αγροτικό και των ε, γεωργικών εργασιών και παροχών ε, αγαθών. Απαντώντας και στον κύριο Λουγιαρίκ, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι πρόθεσή μου να κάνω μία προσαρμογή της κοινή αγροτικής πολιτικής με στόχο να την προσαρμόσω στα αποτελέσματα των διεθνών διαπραγματεύσεων. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Φυσικά έχουν γίνει ήδη τροποποίησεις στην κοινή αγροτική πολιτική για να λάβουμε υπόψη τις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ, διαπραγματεύσεις όπου τα κράτη-μέλη είχαν ήδη ε, εκπροσωπηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τώρα δεν νομίζω ότι είπα ποτέ ότι ένας από τους στόχους της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής είναι να την προσδέσουμε ακόμα περισσότερο στο άρμα των διεθνών διαπραγματεύσεων. Γίνονται αυτές οι διαπραγματεύσεις, έχει καταθέσει μια πρόταση σαφή η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά περιμένουμε να δούμε πώς θα εκτυλιχθεί στο μέλλον αυτή η διαδικασία, αλλά η μεταρρύθμισή μας έχει σαν στόχο να προσαρμόσει τη γεωργία στις ειδικέ ανάγκες και απαιτήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών με τη μεγάλη τη πολυμορφία που είναι το πρόβλημα που αναφέρατε, το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη. Αλλά για το θέμα του εισοδήματο των γεωργών, δεν νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε μια εκπεφρασμένη απάντηση μέσω της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, αλλά μπορούμε να δώσουμε μια, αν θέλετε, ε, υποβόσκουσα ή εγγενή απάντηση. Γιατί εμείς έχουμε σκεφτεί το θέμα του εισοδήματος των διαφόρων κατηγοριών των ε, γεωργών, προσπαθώντας να δούμε πώς θα είναι η κατάλληλη μορφή της απόδοσης αμέσων επιδοτήσεων και ποια θα πρέπει να τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να ανέβουν. Και αυτό είναι μια έμεση απάντηση στο ερώτημά σας. Ανταγωνιστικότητα. Ποια ανταγωνιστικότητα? Είναι κομβικό θέμα. Είναι ένα θέμα που αφορά στην φιλελεύθερη άποψη της γεωργίας και της οικονομίας. Οποιοςδήποτε οικονομικός τομέας πρέπει να αποδείξει ότι είναι φιλελεύθερος και αυτό σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζουμε. Εγώ στην ακρόασή μου είχα αναλύσει το θέμα της ανταγωνιστικότητας λέγοντας ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη διαφορετικότητα των συστημάτων ε, των εκμεταλλεύσεων των χωρών μας και ε, των ε, οικονομικών όρων υπάρχουν ας πούμε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που δεν παράγουν για τη διεθνή αγορά παράγουν για αγορές οι οποίες ε, δεν επηρεάζονται καθόλου από την τιμή των δημητριακών στο χρηματιστήριο του Σικάγου ή του, ή Ρότερνταμ παράγουν για την τοπική αγορά ή μέσα σε ένα σύστημα πολιτικής ποιότητας το οποίο εντάσσεται μέσα, εντάσσεται μέσα σε ένα γενικό ε, ποιοτικό σύστημα. Έχουμε λοιπόν πολλές κοιτίδες παραγωγής που παράγουν ε, μέσα σε ένα πλαίσιο διαφορετικότητας και ως προς το σύστημα παραγωγής αλλά και τις αγορές και την κατανάλωση. Πριν από μερικές εβδομάδε το είπα πάλι στο Κοινοβούλιο ότι η πολιτική ποιότητα είναι ένα σημαντικό σύστημα για το μέλλον της ε, γεωργία και της διαφορετικότητας. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να βρούμε μέσα που θα μας επιτρέψουν να αξιοποιήσουμε αυτή την ανταγωνιστικότητα και τις ιδιομορφίες της και αυτή η ιδιαιτερότητα να γίνει αηφόρος ούτω ώστε ο καταναλωτής να έχει μία σαφέστερη πρόσβαση για το πού θέλουμε να πάμε να προσανατολίσουμε την ΚΑΠ Πού θέλουμε να καταλήξουμε. Δεν θα μακρηγορήσω, θα έχουμε ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Αλλά υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία δεν συνδέονται απόλυτα με μηχανισμούς και πρέπει να το σκεφτούμε το θέμα. Μέχρι τα τέλη της χρονιάς και του χρόνου που θα έρθουμε εδώ με το νομοθετικό πακέτο πάλι θα μιλήσουμε για μηχανισμούς. Αλλά να δούμε πάλι τι θέλουμε για αυτούς τους μηχανισμούς. Ευχαριστώ για όλα όσα μας είπες αγαπητέ Ντάσαν. Συνεχίζουμε. 40 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας. Και με τοποθετήσεις δύο λεπτά το κεφάλι θα μπορέσετε να μιλήσετε όλοι. Ο Τζοβάνι Λαβία έχει το λόγο. Είναι σημαντικός ο ρόλος του στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε για αυτά τα οποία μας είπε σήμερα και θέλω να ευχαριστήσω και τον Τζον Λάιον γιατί η σημαντική του δουλειά αποτελεί σημαντική βάση για συζήτηση. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε ιδιαίτερα σημεία που αφορούν στον προϋπολογισμό. Έτσι όπως φάνηκε σε διάφορες τοποθετήσεις, ο προϋπολογισμός μέσα στο πλαίσιο της ε, η ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΠ παίζει προεξέχοντα ρόλο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η περισχύουσα αρχή του προπολογισμού σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας και η διαπραγμάτευση που κάνουμε ε, με το Συμβούλιο η ψήφο ε, του Κοινοβουλίου είναι αποφασιστική σε περίπτωση διαφωνίας. Για να μιλήσουμε όμως για τα κονδύλια που θα έχουμε στη διάθεσή μας μετά το 2013 για την ΚΑΠ πρέπει να υπογραμμίσουμε το πώς θα διατυπωθεί αυτό το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ήδη ε, με, τη, με την ε, ε, μέση αναθεώρηση Meeting Review στο παλιό δημοσιονομικό πλαίσιο Ξεκινήσαμε τη συζήτηση. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι πια σημαντικό τόσο να μιλήσουμε για το ποια, πόσα θα είναι τα κονδύλια που θα πρέπει, με τα οποία θα πρέπει να πρικοδοτήσουμε την ΚΑΠ. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να πείσουμε το Κοινοβούλιο για τους στόχους της νέας πολιτικής. Δεν πρέπει δηλαδή εμείς να ξεκινήσουμε από τους πόρους για να, πείσουμε το, για να ε, ε, για, να αναπτύξουμε την πολιτική μας, αλλά πρέπει πρώτα να ορίσουμε την πολιτική μας και τους στόχους μας και μετά να ζητήσουμε την πρικοδότηση με τα απαραίτητα ποσά. Εγώ άκουγα πριν τον Κάπουλα Σάντος, ο οποίος μίλαγε για ένα δημοσιονομικό πλαίσιο από τα πριν. Ε, εγώ πιστεύω ότι πρώτα θα πρέπει να ορίσουμε τους στόχους της πολιτικής. Τα κονδύλια θα έρθουν μετά και θα τα ζητήσουμε σε σχέση με τους στόχους. Τώρα, οι αναφορές ε, στην ε, έκθεση του Λάιον. Εγώ θα παρακαλούσα να διαγραφούν αναφορές σε μηχανισμούς, που αφορούν μηχανισμούς και ιδιαιτερότητες του προπολογισμού. Αυτά θα τα συζητήσουμε μετά και θα τα ζητήσουμε μετά, θα τα διεκδικήσουμε μετά, αλλά σε αυτήν την προκατα... προκαταρκτική φάση δεν θα πρέπει να συζητήσουμε αυτά τα στοιχεία. Ινφίνε, εγώ συμμερίζομαι απόλυτα τις θέσεις ε, του Επιτρόπου. Πρώτα πρέπει να μιλήσουμε για τους στόχους της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Θα πρέπει αυτοί οι στόχοι να γίνουν κατανοητοί στους Ευρωπαίους πολίτες. Μετά θα βρούμε τα λεφτά, διότι υπάρχει βούληση στο Κοινοβούλιο. Και όντας το Κοινοβούλιο, βασική αρχή του προϋπολογισμού, θα το πετύχουμε για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τους στόχους που απαιτούν αυτές οι νέες πολιτικές. Ο Στεφάν Λεφόλ. Σε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο που ήρθε εδώ, αλλά και τον George Λάιον. Λοιπόν, πρέπει να αποδείξουμε, κύριε Επίτροπε, ότι η γεωργία έχει ένα ενδιαφέρον για τους πολίτες και πρέπει να γίνει κατανοητή γιατί άμα δεν μας καταλάβουν οι, πολίτες δεν θα μας κατανοήσουν ούτε και οι αρμόδιοι επί του προϋπολογισμού. Πρέπει να έχουμε λοιπόν πολιτικούς στόχους ε, για την ΚΑΠ που να είναι ευανάγνωστοι και κατανοητοί από όλου τους πολίτες διότι αλλιώς θα χάσουμε πολλά. Πρώτο αυτό. Δεύτερο τώρα. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει εμένα είναι να γνωριστεί η διαφορετικότητα των ευρωπαϊκών γεωργιών. Εγώ δεν θέλω να προχωρήσω σε μία εξέγεση της προηγούμενης περίοδου όπου ε, τελικά είχαμε την ε, γεωργία που ήταν ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές και μόνο εκείνη μετρούσε. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη όλους τους τύπους γεωργίας της Ένωσης, διότι αυτό θα έχει επιπτώσεις και στη διαμόρφωση της πολιτικής. Και συγκλίνω τώρα με την έκθεση του George Lyon για το θέμα της αηφορίας της γεωργίας που έρχεται σήμερα στο κέντρο της συζήτησης. Θα έχουμε μια έκθεση στο Στρασβούργο που ελπίζω να υπερψηφιστεί και όπου θεωρείται ότι η Γεωργία αποτελεί λύση για την προστασία της βιοπικιλότητας, των φυσικών πόρων, για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και πιστεύω ότι έτσι οι πολίτες θα μπορέσουν να καταλάβουν και την γεωργική πρόκληση. Για την τροφιμική αυκτάρκεια βεβαίως πρέπει εμείς να έχουμε κατά νου ότι πρέπει να χορτάσουμε τους Ευρωπαίους. 14 εκατομμύρια Ευρωπαίοι υποσυτίζονται σήμερα και πρέπει να τους καλύψουμε. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να μπουν επιτάπητος. Και οι γεωργικές και τροφιμικές πολιτικές πρέπει να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτηματικά. Όπως είπε και ο Τζόρτζ στην έκθεσή του, εγώ θα έδινα τρεις βασικούς στόχους και προκλήσεις για την ΚΑΠ. Πρώτον, ρύθμιση των αγορών. Και στην έκθεση του George Lyon απέχουμε παρασάγκας από το να μιλήσουμε για οργάνωση αγορών και, έχουμε, και εξού δηλαδή και όλο αυτό το σκαμπανέβασμα των τιμών. Δεύτερον, αντιστάθμιση όλων των handicap, όλων των προβλημάτων. Δηλαδή, οι αποζημιώσεις και αντισταθμίσεις να μην χρηματοδοτούνται μόνο από τον δημόσιο τομέα. Τρίτο, είπαμε ρύθμιση, αποζημιώσεις και πληρωμή των υπηρεσιών και κλίμα. Θεωρώ λοιπόν ότι η συζήτηση σε καλή βάση, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε μακρύτερα, διότι αλλιώ εμεί δεν θα απαντήσουμε στι προσδοκίε των γεωργών, κυρίω με την κρίση που του πλήττει σήμερα και για το γάλα, αλλά αυτή η κρίση σήμερα προχωράει και πλήττει άλλου τομεί, ε, τα δημητριακά και άλλους. Αυτά βέβαια πρώτα πρέπει να τα συζητήσουμε μεταξύ μας και θα ολοκληρώσω τώρα με τα διεθνή. πρέπει να το πούμε στην Επιτροπή Γεωργίας σαφέστατα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να έχει ως διαπραγματευτική στρατηγική το άνοιγμα των γεωργικών αγορών όταν η ίδια θέλει να προωθήσει βιομηχανία και υπηρεσίες στον κόσμο. Δεν είναι μόνο πρόβλημα της ΠΟΕ, είναι το πρόβλημα το πώς εμείς διαπραγματευόμαστε σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό γίνεται πάντα εις βάρος της γεωργίας και του, του, του προβλήματος. Αυτό πρέπει να το πούμε, δηλαδή άμα θέλουμε να μετρήσουμε διεθνώς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε για την ευκαιρία που μας δίδεται να συζητήσουμε για το θέμα αυτό και να ξεκινήσουμε μια συζήτηση η οποία θα καλύψει όλη την κοινωνία μας. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Λάιον γιατί η έκθεσή του με, με πολύ θετικό τρόπο αντιμετωπίζει όλη αυτή την προβληματική. Θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο μας λένε πάντα οι γεωργοί όταν συναντιόνται μαζί μας. Θέλουν να ξαναγίνουν ανταγωνιστικοί. Θέλουν εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πιέσουμε την Κομισιόν και το Συμβούλιο να αρθούν οι φραγμοί που τους επιτρέπουν να ανταγωνιστούν με ισότητα μέσα σε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς όπως έχουμε στην Ευρώπη. Για να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικοί πρέπει να λύσουμε πολλά προβλήματα, κατά από τα οποία έχουν αναφερθεί ήδη σήμερα το απόγευμα. Δηλαδή, ποια θα είναι τα μέτρα, παραδείγματο χάρη, τα οποία θα δώσουν στους παραγωγούς τη δυνατότητα να έχουν διαπραγματευτική θέση μέσα στην τροφιμική αλυσίδα και να αποφευχθούν οι καταχρήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή. Πώς θα αντιμετωπιστεί η υπερβολική διακύμανση των αγροτικών τιμών. Θεωρεί ο κύριος Επίτροπος ότι είναι δυνατόν μέσα στα πλαίσια της, του ΠΟΕ να υποστηριχθεί η αρχή της αμοιβαιότητας σε ό,τι αφορά την ευζοία των ζώων, το περιβάλλον και η τροφιμική ασφάλεια. Ένα τελευταίο θέμα ενώπιον των διαπραγματεύσεων με τρίτε χώρε για διμερεί συμφωνίε, παραδείγματο χάρη, όπω έχουμε κάνει με το Μαρόκο, εμεί διαπιστώσαμε ότι δεν, συμπληρω... συμπεριλαμβάνουν κάποιο μηχανισμό που θα εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με αυτό το μηχανισμό από την πλευρά τρίτων χωρών. Ξέρουμε ότι υπάρχουν συστηματικέ παραβιάσει. Υπάρχει κάποιο μέτρο το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να εισαχθεί ώστε οι τρίτε χώρε να εκπληρούν αυτά τα οποία υπογράφουν στι συμφωνίε μαζί μα. Γιατί είναι σαφέ ότι η παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σέβονται μέχρι κεραίας όλα αυτά τα οποία του ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, ποιος θα είναι ο ρόλος της διαμόρφωσης μετά το 2013. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε για χρήματα αυτή τη στιγμή, αλλά αν επανέλθουμε στα χρηματικά, θα πρέπει ίσως να επανέλθουμε στην ε, διαμόρφωση σαν λύση για τους γεωργούς ενώπιον της τσιγκουνιάς των κρατών μελιών. Ο Μάρκ Θεραμπέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ευχ... Σας ε, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Και χαιρετίζω το γεγονός ότι δεν είστε επίτροπος της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, αλλά των Ευρωπαϊκών Γεωργιών, και ότι πολύ σωστά το δάσος εκφράζει πιο πλουραλιστικά το δέντρο. Ο Γιωργός ε, είναι παραγωγός ε, κοινή ωφελία. Αγαθών κοινή ωφελία. Θέλουμε επίσης, όπως λέει η έκθεση, μία πιο αηφόρο, κάπ, ε, και όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Τώρα στην παράγραφο 19 ο George Λάιον αναφέρει για τις διάφορες για τα διάφορα προβλήματα των αγορών όπως η αστάθεια των τιμών κλπ. Και δεν έχουμε λύση. Και κύριε Επίτροπε, εγώ να σας πω και χαίρομαι για αυτά που είπατε για το γάλα. Ότι δεν περιμένετε το 2013 για να αντιδράσετε το γάλα. Είναι ένας τομέας που όπως το δέντρο κρύβει και άλλους τομείς. Διότι και τα δημητριακά πλήττονται από την αστάθεια και τα κρέατα Μην μας τα πείτε βέβαια σήμερα, δεν είναι αυτός ο στόχος. Αλλά τέλος πάντων εσείς ε, θα μπορούσατε να παίξετε ένα ρυθμιστικό ρόλο ε, και να ορίσετε και την ε, δυναμικά, τον, τη δημόσια άποψη για όλα αυτά. Βεβαίως δεν είμαστε στη Στρέσα ούτε και στους υπουργούς που ήταν τότε εκεί και υπερασπιζόταν αυτά τα ιδανικά. Αλλά τέλος πάντων σήμερα πώς μπορούμε εμείς να προστατεύσουμε τους αγρότες και τις αγρότησες. Και θέλω να σας ακούσω κύριε Επίτροπε να μου πείτε εσείς ε, τι ρόλο θα παίξετε ως ε, ρυθμιστικό στοιχείο στην αγορά και πώς θα επιτρέψετε και στο δημόσιο χώρο να παίξει το ρόλο του. Ο κύριος Μποβέ Και εγώ θέλω να παρεμβώ μετά από αυτά τα οποία ελέγχθησαν από τον κύριο Επίτροπο και φυσικά από αυτά που είπε ο κύριος εισηγητής. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό είναι ότι υπάρχει η θέληση να υπάρχει μια συνολική αντιμετώπιση, μια αντιμετώπιση που στρέφεται προς το μέλλον. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει όμως συγχρόνως να προσέξουμε να μην ξανακάνουμε αυτό που είχαμε κάνει το 1991 με την έκθεση Μαξάρι η οποία είχε αντιμετωπιστεί και φαντα... την είχαν δει πολύ σαν μια πραγματική τομή για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η πολιτική υπέρ των γεωργών. Γιατί τα αποτελέσματα αυτής της πρότασης ήταν ακριβώς αντίθετα από τις ελπίδες που απεδείχθησαν φρούδες της πρότασης Μαξάρι. Και είδα ότι υπήρξε πραγματικά εξέγερση και μεγάλη απογοήτευση στον αγροτικό κόσμο. Γι' αυτό λέω ναι, μια σημαντική συζήτηση θα πρέπει οι πολίτες να συμμετάσχουν και φυσικά και οι οργανώσεις των παραγωγών, αλλά αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία όλης αυτής της διαδικασίας, θα πρέπει τα εργαλεία τα οποία θα προέρθουν από αυτήν την συζήτηση να αναπτύξουν, να αναπτυχθούν μάλλον μέσα στο πλαίσιο του πνεύματος μέσα στον οποίο θα γίνει η διαβούλευση. Να γυρίσουμε στο 1954 να θυμηθούμε ποιο ήταν το πνεύμα της κοινή αγροτικής πολιτικής, γιατί κανένα δεν το είπε αυτό. Ήταν το πρώτο εργαλείο για να εξασφαλίσουμε την ειρήνη στην Ευρώπη. Ήταν ένα κεντρικό θέμα. Το θέμα της ειρήνης και της τροφιμικής και γεωρικής πολιτικής. Να μιλάμε για γεωρική και τροφιμική πολιτική λοιπόν και τα δύο μαζί ως στοιχείο ειρήνης συνοχής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 μελών σήμερα, αλλά επίση και κάτι που αποτελεί στοιχείο συνεκτικό σε σχέση με τον έξω χώρο. Γιατί σήμερα αυτό το οποίο αναμένουν <clears throat> οι χώρες, οι τρίτες χώρες και ιδίως οι χώρες του τρίτου κόσμου του Νότου είναι η ευρωπαϊκή πολιτική γεωργίας να μην στρέφεται κατά της ανάπτυξης των δικών τους γεωργιών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να διαθρέψει τους, Ευρώπους με, τους Ευρωπαίους με υψηλό επίπεδο και με προστασία του περιβάλλοντος και με διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, αλλά δεν πρέπει να έχει αντικό αντίκτυπο έξω από την Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν μια συνένεση και είναι κεντρικό εδώ το θέμα της επίπτωσης στη γεωργία του τρίτου κόσμου. Έχουμε τώρα ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι οι συμφωνίες του ΠΟΕ με τη μορφή που έχουν παρουσιαστεί και από πολλούς προλαλήσαντες. Όχι γιατί μονάχα θα πρέπει να υπάρχει κατάργηση αυτών των συμφωνιών. Πρέπει να υπάρξουν συμφωνίες αλλά από τη βάση νέων στοιχείων. Ένα βασικό στοιχείο συνδέει σήμερα την κοινή αγροτική πολιτική με, τη, με τον ΠΟΕ που είναι το θέμα των διεθνών τιμών. Οι τιμές που έχουμε στην Ευρώπη για τα τροφιμικά προϊόντα είναι οι διεθνείς τιμές. Αλλά όλοι ξέρουν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν ότι αυτές οι τιμές είναι γαργαλημένες, δεν καμία οικονομική σημασία είναι τιμές dumping και όχι τιμές παραγωγής ούτε για τους Ευρωπαίους γεωργούς ούτε για τους γεωργούς του άλλου κόσμου. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να λάβουμε υπόψη αυτό το στοιχείο και να εξασφαλίσουμε μια δικαιοσύνη, όχι μόνο μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε διεθνές επίπεδο να αποκαταστήσουμε τις πραγματικές τιμές. Και εδώ επανέρχομαι στο θέμα της ε, ειρήνης και της ανάγκης να έχουμε μια πολιτική ειρήνη σε παγκόσμιο επίπεδο. Τελευταίο στοιχείο. Κάτι ακόμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Ένα ερώτημα το οποίο δεν αναφέρθηκε στον κατάλογο των, ε, ε, του κύριου Επιτρόπου είναι το θέμα της πρόσβασης στη γη και της διατήρησης της ποιότητας των γεών για τις επερχόμενες γενναίες. Θα πρέπει η Ευρώπη να δώσει δυνατότητα στους νέους που εγκαθίστανται στη γεωργία να έχουν πρόσβαση στην ε, αγροτική γη, παρά την πολυπλοκότητα των συστημάτων αγροτικής ε, ιδιοκτησίας στα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να προστατεύσουμε και αυτές τις γης ενώπιον της ε, κερδοσκοπίας που γίνεται πολλές φορές. Για να μιλήσουν όλοι θα πρέπει να επιταχύνουμε λιγάκι. Ο κύριος Σταμπάτζη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, έχετε μεγάλο δίκιο όταν λέτε ότι πρέπει να πείσουμε τους φορολογούμενους. Αποκλίνουν όμως πολύ τα επιχειρήματά μας. Δεν υπάρχει μια ικανοποιητική σύγκληση των επιχειρημάτων σε σχέση με το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής. Παραδείγματος χάριν, η αγορά των δημοσίων, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αγαθών. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό επιχείρημα αλλά δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ποσοτικοί υπολογισμοί ούτε καν κατά προσέγγιση για το ποιο είναι το κέρδος που αποκομίζει η κοινωνία μας από τα δημόσια αυτά αγαθά που παράγουν οι γεωργοί και οι εργαζόμενοι στον αγροτικό χώρο. Οι αγορές λοιπόν δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τον τρόπο αυτό, χωρίς να ξέρουμε το κόστος αυτών των αγαθών των κοινωνικών και περιβαλλοντικών. Αγαπητοί συνάδελφοι, εξάλλου δε, στην πρώτη μορφή που είχε λάβει η στατηγική 2020, δεν υπήρχε η παραμικρή αναφορά στην κοινή αγροτική πολιτική. Θα πρέπει λοιπόν να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Μπαρόζο, καθώς και τους Υπουργούς Οικονομικών, να εξασφαλίσουμε μια σύνδεση των στόχων μας στην κοινή γεωργική πολιτική, με την πράσινη πολιτική, με την καινοτομία, με τους νέους στόχους που αφιδώς έχει διατυπώσει ο κύριος Παρόσο για το 2020. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Υπάρχει και ένα περαιτέρω θέμα, κύριε Επίτροπε, το να μπορέσουν να προλάβουν οι νέες χώρες μέλη τις παλιές. Μιλήσατε για την πολυμορφία των 27 χωρών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα γεωργίας. Αλλά μέχρι το 2013 οι χώρες που έχουν μπει πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι σε θέση να προλάβουν τις παλιές χώρες. Μήπως θα υπάρχουν κάποιες, κάποια μέσα για να το πετύχουν αυτό στη συνέχεια. Και ένα συγκεκριμένο ερώτημα, κύριε Επίτροπε, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά το moratorium για την αγορά από το εξωτερικό προϊόντων από τα νέα κρατημέλη. Αν τα νέα κρατημέλη δεν πάρουν μια παράταση της απαγόρευσης αυτής, θα υπάρξουν τεράστιες διαταράξεις στην αγορά των νέων κρατών μελών. Γιατί γίνεται από την πλευρά της Κομισιόν μια τέτοια προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εγώ είμαι στην ακατανοησία σε σχέση με τη λογική. Μουλτσουμές και σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ντελάνζ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Επίτροπο που ήρθε και μετά να συγχαρώ τον συνάδελφο για την έκθεσή του. Τα βασικά στοιχεία περιέχονται και συμφωνώ πως ε, με τον πρώτο μιλητή των Πρασίνων πως ε, είναι κάπως υπερσιόδοξο το ότι η κυνηγερική πολιτική επέτυχε τους στόχους για ένα δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες. Ίσως να ήταν έτσι κάπως ε, υπερβολικό αυτό το συμπέρασμα. Κάποιες παρατηρήσεις. Τώρα για μια φιλελεύθερη καινοτομία εμφανίζεται λίγο αργά στην ε, έκθεση, ίσως για τους Ολλανδούς φιλελεύθερους. Εμεί θα το βάζαμε οπωσδήποτε πιο νωρί και να γίνω πιο συγκεκριμένη για το ζήτημα τη κλιματική αλλαγή. Ε, πολύ σωστά υπογραμμίζεται τον ρόλο του εδάφους όταν μιλάμε για τη δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα και τη μείωση των εκπομπών, αλλά νομίζω πως είναι πολύ περιορισμένο γιατί και οι γεωργικοί τομείς που δεν έχουν πολύ έδαφος, π.χ. οι εντατικοί τομείς έχουν να παίξουν μεγάλο ρόλο όταν μιλάμε για τη μείωση των εκπομπών. Μιλάμε εδώ πέρα για τα θερμοκήπια της Ολλανδίας παραδείγματο χάρη, Οπότε με την άδειά σας θα ήθελα να διευρυνθεί αυτό το κομμάτι εδώ πέρα για να συμπεριληφθούν και άλλοι τομείς. Συμφωνώ επίσης ε, για το θέμα των αντικειμενικών κριτηρίων που χρειάζονται για να ε, ορίσουμε τις ε, πληρωμές. Επίσης αγοραστική δύναμη ενδιαφέρον, το κόστος γενικότερα και θα ζητήσω και πάλι από την Κομισιόν. Αυτό το κάνω κάθε φορά που το συζητάμε αυτό το θέμα. Ζητάω, ρωτάω την Κομισιόν τι γίνεται με τα πιλωτικά έργα που ζητήσαμε πριν από λίγα χρόνια στον προϋπολογισμό λέμε δείτε λίγο κάποια αντικειμενικά κριτήρια για να χρησιμοποιήσουμε. Γνωρίζουμε πως θα γινόταν αυτή η συζήτηση. ζητήσαμε μια μελέτη ή έργα και κάθε φορά που λέω κάτω από την Κομισιόν με κοιτούν πανικόβλητοι. Και ε, κάθε φορά μου λένε θα το δούμε και θα σας πούμε. Ελπίζω αυτή τη φορά η Κομισιόν να έχει κάτι να μου πει και δεν θα μου πει πάλι ότι θα το δει και θα με ειδοποιήσει. Δύο διευκρινήσεις ε, για τον εισηγητή, δύο Είπατε πώς θα πρέπει η κοινή γεωρική πολιτική να ενταχθεί σε μια πολυλειτουργική πολιτική τροφίμων. Τι σημαίνει αυτό, ποια άλλα στοιχεία θα έχει αυτή η πολιτική τροφίμων ή θέλετε να αντικαταστήσετε την γεωρική πολιτική από μια πολιτική τροφίμων. Δεν έχω καταλάβει. Και τελευταία ερώτηση, όταν φύγουμε από τις ιστορικές πληρωμές, αναφέρατε το πρόβλημα της γυμνής γης. Δεν θα προσπαθήσω καν να το μεταφράσω, αλλά νομίζω πως έχουμε το, το αντίστοιχο πρόβλημα στο δικό σας κρατός μέλος, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εάν φύγουμε από τις ιστορικές πληρωμές, ξαφνικά υπάρχει μια μεγάλη αύξηση στις αιτήσει ε, για ενιαία πληρωμή, γιατί κάθε πλούσιος οδοντίατρος που έχει εκεί πέρα ένα χωραφάκι και δύο πόνι ε, ζητά επιδότηση. Ε, δεν παράγει τρόφιμα βεβαίως αυτός ο άνθρωπος, οπότε πώς θα φύγουμε από τις ιστορικές πληρωμές, αλλά να παραμείνουν οι πληρωμές κατά κάποιον τρόπο συνδεδεμένες με την παραγωγή τροφίμων. Γιατί όταν μιλάμε νομίζω για ασφάλεια τροφίμων, αυτό είναι το βασικό. Σας ευχαριστώ κύριο Σμιτ. Ελπίζω να καταφέρετε να κρατήσετε το χρόνο σας γιατί αλλιώς δεν θα πάρουν το λόγο οι τελευταίοι τρεις εγγεγραμμένοι. Ναι, θα είμαι σύντομος γιατί μπορώ να συγχαρώ τον συνάδελφο, συνάδελφο ενό Σκοτσέζο, δεν είμαστε στην ίδια ομάδα, τον ε, εισηγητή, τον κύριο Λάιον και συμπατριώτη δηλαδή. Και κάτι το οποίο δεν ανέφερε κανείς και μου απογοητεύει λίγο, η Επιτροπή Ανάπτυξης δεν μας έδωσε γνωμοδότηση εδώ πέρα και οπωσδήποτε νομίζω είναι θεμελιώδης η μετάρρυθμιση κοινής γεωρικής πολιτικής για την ανάπτυξη. Και ίσως εσείς οι συντονιστές θα μπορούσατε να το ζητήσετε να το ξαναδούν, γιατί οπωσδήποτε θέλουμε συνεισφορά από αυτή την Επιτροπή. Επίσης για τις μειονεκτικές περιοχές νομίζω δεν μπορούμε να το τονίσουμε αρκετά. Είναι ένα κομμάτι που νομίζω πάρα πολύ καλά αντισταθμίζει τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από την γεωργική πολιτική. Νομίζω ο Τζόρτζ το ξέρει πως θα πρέπει, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τη λήψη αποφάσεων σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς ε, Εθνική Αρχή δεν σημαίνει οπωσδήποτε το κράτος μέλος. Επίσης, ε, ενεργή γεωργία, το ορισμός το είδαμε πολλές φορές. Ε, πιέζεται ο προπολογισμό, ε, ο γεωργικός, αυξάνεται ο παγκόσμιος πληθυσμό, έχουμε την κλιματική αλλαγή, δεν μπορούμε να στηρίζουμε δραστηριότητες που δεν είναι παραγωγή τροφίμων. Πρέπει η κοινή γεωργική πολιτική να αφορά την παραγωγή τροφίμων, αλλιώς θα δούμε πως θα έχουμε άσχημα αποτελέσματα, αναποτελεσματική χρήση των δημοσίων κονδυλίων. Οπότε δέντρα πτηνά τα οποία δεν είναι παραγωγικά, καπνά κτλ. Μπορεί να είναι γεωργική δραστηριότητα, δεν εμπίπτουν στην ε, κοινή γεωργική πολιτική. Επίση, ανησυχώ πω τελικά θα καταλήξουμε, δεν θα κάνουμε τίποτα. Πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Υφίσταται φοβερή πίεση ο υπερπολογισμό. Και αν βάζουμε στόχο και στόχο και στόχο και στόχο, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα, δεν θα κάνουμε τίποτα. Υπάρχει κίνδυνο εδώ πέρα πω η Γενική Διεύθυνση Γεωργία εδώ πέρα έχει τόσο τομεί ε, πολιτική και δεν υπερασπίζεται τον ίδιο τον προπολογισμό τη. Ε, και εδώ πέρα έχουμε το θέμα τη πράσινη ανάπτυξη. Πρέπει και εμεί να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Πρέπει να πάμε στα διαρθρωτικά ταμεία για αυτό το θέμα, αντί να πάνε τα κονδύλια τη κοινή γεωργική πολιτική και να διαμεριστούν ακόμη περισσότερα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ για την επίσκεψή σας. Ευχαριστώ και τον εισηγητή που είμαστε το έγγραφο. Αναφέρομαι σε αυτά τα οποία και είπατε και σήμερα αλλά και άλλες φορές. Θέλω να πω ότι ακούμε και ξανακούμε σε αυτή την αίθουσα πρέπει, πρέπει και πρέπει. Ε, εσείς όμως προσθέσατε όμως κάτι καινούργιο. Ναι, πρέπει να κάνουμε κάτι, αλλά πώς. Και αυτό πρέπει να πούμε και στους Γιωργούς που περιμένουν απαντήσεις ε, στις ερωτήσεις μας. και ελπίζω ότι εσείς θα μπορέσετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας, όχι μόνο τις δικές μας αλλά και των αγροτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν στη διάθεσή τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι, έχουν όλα τα μέσα και τις δυνατότητες να εργαστούν σωστά αυτοί λοιπόν πρέπει να προτείνουν τις λύσεις. Χρειάζεται να έχουμε επαφή με τους γιοργούς. Δεν πρέπει να περιμένουμε οι μπαμπάδες μας ή οι παππούδες μας να μας πούνε ποια θα είναι τα μέτρα που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και ξανά πρέπει. Αλλά πώς να αλλάξουμε... Εσείς είπατε σήμερα ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μία ανακατανομή των πληρωμών για να πετύχουμε ισοτιμία. Πώς θα το κάνουμε όμως αυτό? Με έναν ειδικό προϋπολογισμό. Εμείς δεν θέλουμε έναν πιο περιορισμένο προϋπολογισμό από αυτόν που έχουμε και η συγκεκριμένη ερώτηση πώς θα μοιράσουμε εμείς αυτές τις πληρωμές βάσει εκταρίων υποστηρίζοντας όμως παράλληλα και τους βιολογικούς καλλιεργητές. Ήρθε λοιπόν η ώρα να συζητήσουμε και τις εφαρμοστικές λεπτομέρειες όλων αυτών των πραγμάτων. Σε αυτή την αίθουσα έχουμε ακούσει πολιτικούς εμπειρογνώμονες να μιλάνε για προϋπολογισμό. Γνωρίζουμε την ε, γεωργία, όχι, όλη τη γεωργία, όχι μόνο τη γεωργία, τη βιομηχανική γεωργία, την ε, γεωργία ως business. Εμείς διατρέχουμε τον κίνδυνο να σπαταλήσουμε τον προϋπολογισμό. Πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα όμως τα υπάρχοντα κονδύλια Θα ήθελα λοιπόν να μην μιλάμε μόνο για έναν γενικό προϋπολογισμό, αλλά το πώς θα αξιοποιήσουμε αποτελεσματικότερα τον προϋπολογισμό που έχουμε. Σίγουρα πρέπει να μιλήσουμε για μια αναδιανομή των πληρωμών στην ΚΑΠ. Ως ένα βαθμό έχει γίνει αυτή η ανακατανομή, αλλά πρέπει να βρούμε ποιος είναι ο σωστότερος δρόμος. Διότι δεν φτάνει να ζητάμε μόνο έναν παχύ προϋπολογισμό, διότι αυτός ο προϋπολογισμός δεν θα λύσει το πρόβλημα του πώς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ε, κύριε Επίτροπε, για την ε, παρουσία σας ε, σε αυτή την Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει θα γυρίσω στα αγγλικά για να με ακούσετε και να απαντήσετε. Εγώ συναντώ πολλούς λετωνούς αγρότες και θα τους ενημερώσω και για τις συζητήσεις μας. Πρώτα απ' όλα οι λετωνοί αγρότες καλωσορίζουν την συνένεση για το ότι η άμεση στήριξη στους αγρότες πρέπει να φύγει από το σύστημα το ιστορικό και να πάει σε ένα σύστημα σε αντικειμενικά κριτήρια. Αλλά παραμένει το ερώτημα. Αντιμετωπίζουμε ακόμα μία περίοδο μέχρι το 2020 προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα. Όπως γνωρίζετε, οι αγρότες και οι πολίτες, όχι μόνο στη Λετωνία, σε όλα τα νέα κράτη-μέλη ε, που λαμβάνουν πολύ λιγότερες άμεσες πληρωμές δεν συμφωνούν με αυτή την ε, μεταβατική περίοδο. Θυμούνται πως δεν υπάρχει ουδέν ε, μονιμότερον του προσωρινού και επανειλημμένα έχουν ζητήσει δίκαιη και ίση μεταχείριση όλων των γεωργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την επόμενη περίοδο του προπολογισμού. Και αυτό δεν είναι ζήτημα περισσότερων άμεσων πληρωμών, είναι ζήτημα ίση μεταχείρισης σε ένα δίκαιο σύστημα. Ακόμα και αν αυτό σε απόλυτου αριθμού είναι μικρότερο ποσό. Είναι ζήτημα δίκαιου ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, ε, παρά ζήτημα του να λάβουν περισσότερα χρήματα. Εγώ όμως είμαι πολιτικός και εμείς οι πολιτικοί αντιλαμβανόμαστε πως καμία πολιτική, ειδικά τόσο σημαντική, δεν μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία οποιαδήποτε μεταβατική περίοδος να οδηγήσει σε ένα δίκαιο σύστημα το οποίο θα οδηγήσει σε μια Ευρώπη ε, των πολλών ταχυτήτων, την οποία θα στηρίζουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Επίσης, οι αγρότες στη Λετωνία καλωσορίζουν το ότι δεν θα επιστρέψουμε στις συνδεδεμένες πληρωμές. Λένε πως η αλλαγή θα πρέπει να είναι συνολική, όλη η άμεση στήριξη θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την παραγωγή χωρίς εθνική σχηματοδότηση και χωρίς εξαιρέσεις. Και Καταλήγοντα, επίση πιστεύουν οι αγρότε στη χώρα μου πω αρχή τη διάρθρωση δεν θα πρέπει να αποτελέσει μέλο της μελλοντική ε, ΚΑΠ γιατί υποβαθμίζει και υπονομεύει την δικαιοσύνη μεταξύ αγωτών σε διαφορετικές περιοχές και κράτη-μέλη. και μετά Γκαρσία Πέρες. Λοιπόν, σεβαστείτε το χρόνο σας, αλλιώς δεν τα καταφέρουμε. Uh, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι για το γεγονός ότι πιστεύετε σε μια ισχυρή και νεαγροτική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Γεωργία και προφανώς και ένας εύρωστος προϋπολογισμός είναι απαραίτητο για να γίνει αυτό. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα σε σχέση με τις γαλακτοκομικές ποσοστώσεις. Πολλοί γεωργοί στη Βόρεια Ελλάδια από όπου έρχομαι έχουν αντιμετωπίσει μεγάλη πίεση στο γαλακτοκομικό τομέα. Στην Βόρεια Ελλανδία τον τελευταίο καιρό έχουμε δει να είναι χαμηλότερες τιμές από ό,τι ήταν ποτέ στη ζωή μας. Και επομένως, από αυτά που είπατε καταλαβαίνω ότι χρειάζεται, ότι συμφωνείτε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν μέτρα για την αντιμετώπιση της αστάθειας των τιμών στην αγορά. Θα ήθελα όμως να υπάρξει άμεση δράση σε σχέση με το γαλακτοκομικό τομέα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολλοί γεωργοί οι οποίοι δεν μπορούν να συνεχίσουν με αυτού του ταχύ κύκλου ανάπτυξη και κατάρρευση και δεν έχει κανένα νόημα να μιλάμε για μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτική, εάν δεν θα υπάρχουν πια αυτοί οι γεωργοί να ωφεληθούν από αυτή την μεταρρύθμιση. Και αν μπορώ τώρα να σταθώ στην έκθεση του Γεωργίου Λάιον, να τον ευχαριστήσω για την έκθεσή του. Η έκθεσή του είναι αξιο... αξιέπαινη, θέτει πάλι όμως ορισμένα ζητήματα που φέρνουν μεγάλη αβεβαιότητα για τους γεωργούς στη Βόρεια Ιρλανδία. Οποιαδήποτε καταποκοπή σε σχέση με την ε, έκταση μονάχα επιδότηση θα έχει μεγάλη επίπτωση για τους γεωργούς στην ε, Βόρεια Ιρλανδία. Ένα από τα σημαντικά θέματα είναι το πώς θα συνδέσουμε την κοινή γεωργική πολιτική με την παραγωγή τροφίμων και όχι μονάχα με τη χρησιμοποίηση της γης. Δεν θέλουμε επίσης να υπάρξει συγχρηματοδότηση γιατί θα δημιουργήσει ίσως πολλά προβλήματα και θα δημιουργήσει και άνισε συνθήκες ανταγωνισμού για πολλούς από τους γεωργούς που προσωπώ σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Όπως λέμε και στη Βόρεια Ιρλανδία, ο διάβολος είναι στις λεπτομέρειες. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μια συζήτηση η οποία πρέπει να λάβει χώρα, όχι μόνο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων για όλα αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Γκαρσία Περές και μετά Μαγκίνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, Επίτροπο και τον συνάδελφο Λάιον. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που έχουμε σήμερα και πιστεύω ότι πρέπει να είναι μία συζήτηση όπου συνειδητά αναγνωρίζεται η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα στο γεωργικό τομέα στην Ευρώπη. Μιλάμε για κρίση και πρέπει να, έχουμε, να συνειδητοποιούμε ότι οι αγρότες προσδοκούν από τα ευρωπαϊκά όργανα, κομισιόν, κοινοβούλιο, ότι είμαστε ικανοί να απαντήσουμε στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας προκλήσεις που μπορέσαμε ήδη να τις ε, δούμε ποιες είναι, να τις διαπιστώσουμε και υπάρχει μια γενική συμφωνία γύρω από όλα αυτά, τροφιμική ασφάλεια, ε, θέση εργασίας στην Ήπεθρο, συνεισφορά της ε, γεωργίας στον αγώνα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να δούμε τώρα πώς θα απαντήσουμε σε όλα αυτά και να δώσουμε ασφάλεια στους ε, Ευρωπαίους αγρότες. Διότι υπάρχει μια τεράστια αβεβαιότητα όπως σας είπα σχετικά με τις άμεσες πληρωμές. Πρέπει να είμαστε σαφείς για το πώς μέσα από τη νέα προπτική που θα ξεκινήσει με τη νέα ΚΑΠ το 2013 θα μπορέσουμε να απαντήσουμε και με μέτρα διαχείρισης των αγορών και πώς αυτές οι αγορές θα είναι οργανωμένες κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ παραγωγής και εμπορίας. Πρέπει να δούμε πώς θα απαντήσουμε στην κατάσταση μια μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων πρωταγωνιστών που συμμετέχουν στην τροφιμική αλυσίδα. Και θέλω να απαντήσω, στον, να, να, να, να ρωτήσω τον Επίτροπο. Μιλήσατε για τη στρατηγική 2020 και έγινε αναφορά στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σε μία από τις παραγράφους λέει το πώς η νέα ΚΑΠ μπορεί να συμβάλλει στην προσέγγιση των στόχων του 2020. Μιλάμε λοιπόν για τη γεωργία ως στρατηγικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα απαντήσει λοιπόν στους στόχους της 2020 η γεωργική πολιτική. Μαγκίνες. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο και τον εισηγητή για τη σημερινή συζήτηση η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα οπωσδήποτε αλλά εγώ αν ήμουν αγρότης θα έκανα το βασικό ερώτημα. Δίνει κατευθύνσεις στους αγρότες για το τι πρέπει να κάνουν και δεν το κάνει αυτό και νομίζω το μήνυμα σήμερα προς τους αγρότες εάν ακούνε είναι πως δεν υπάρχει σαφήνεια εδώ πέρα και ο Επίτροπος λέει πως σωστά θα πρέπει να σπεύσουμε βραδέως και να δούμε όλες μας επιλογές ε, για το έγγραφο για τη δημόσια διαβούλευση. Το καλωσορίζουμε, αλλά εμένα μου φοβίζει πολύ η δημόσια διαβούλευση χωρίς κατευθύνσεις, γιατί πρέπει να ενημερώνονται οι άνθρωποι πριν ε, ε, λάβουν μέρος σε μια συζήτηση. Και Νομίζω πως οι Ευρωπαίοι καταναλωτές ε, θέλουν τα υψηλά ποιοτικά τρόφιμα και αντιλαμβάνονται τα προβλήματα των αγροτών. Οπότε ενδιαφέρον θα είναι να δούμε το τι θα προκύψει από την διαβούλευση. Εγώ θα ήθελα η Κομισιόν να έχει καλύτερα μέσα πρόβλεψης του μέλλοντος. Γιατί όσον αφορά τις τελευταίες αυξήσεις και μειώσεις τιμών δεν τα πήγαν πολύ καλά οι ειδικοί. Επίσης, θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιό να επανέλθει κάποια άλλη ημέρα για το όταν θα έρθει στην επικαιρότητα αυτό το θέμα αργότερο, αργότερα εντός του έτους για το ποιος λαμβάνει ποια επιδότηση και αυτό αφορά πάρα πολύ τα μέσα. Εάν αλλάξουμε και πάμε σε ένα σύστημα πληρωμής για κάποια δημόσια αγαθά πάλι η ίδια κατανομή δεν θα είναι. Γιατί ε, φυσικά βεβαίως η μεγάλη παραγωγή τώρα λαμβάνουν τι μεγάλες ε, πληρωμές λόγω του όγκου της παραγωγής και οπωσδήποτε όσοι έχουν μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις θα ε, προσφέρουν περισσότερα δημόσια αγαθά και θα έχουν περισσότερες πληρωμές. Μπορεί να μας το αναλύσει αυτό η Κομισιόν, πώς κατανέμονται οι πληρωμές με το κάθε διαφορετικό σενάριο. Επίσης να περάσω στην πολύ καλή έκθεση του George Lyon, που χαίρομαι που δεν είναι πολύ συγκεκριμένη αλλά οπωσδήποτε είναι κάποιες, ε, δίνει κάποιες καλές αρχές. Τώρα για τον προπολογισμό, η παράγραφος 45 μιλάει για διατήρηση του προπολογισμού και η 57 και 59 νομίζω πως μιλάνε για αύξηση του προπολογισμού για άλλα μέτρα. Θα πρέπει ίσως να το δούμε αυτό. Παράγραφο 60 για τα βιοκαύσιμα και βιοαπόβλητα. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρονται τα κράτη-μέλη και νομίζω και εμεί δεν ξέρουμε τι κάνουμε εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να είμαστε σαφεί όσον αφορά τους αγρότες που το χρειάζονται. Και επειδή βεβαίω ε, και ο χρόνο έχει τελειώσει, πρέπει να καταλάβουμε πω οι αγρότε δεν πληρώνονται δίκαια για την παραγωγή του. Εάν δεν το πληρώνουν οι πρέπει να πληρωθεί με έναν άλλο τρόπο και πρέπει να βρούμε το μηχανισμό. Και τέλος, ανησυχώ για την λέξη πράσινη. Το πράσινος έχει γίνει το νέο χρυσός και ό,τι γυαλίζει δεν είναι χρυσός, ό,τι είναι πράσινο δεν είναι καλό. Κάμια φορά έχουμε λάβει πράσινες πρωτοβουλίες και είχαμε λάθος αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δανέλης, μετά Ανιό και για ένα λεπτό, αλλιώς δεν θα τα καταφέρουμε να κλείσουμε. Θα αναφερθώ σε ένα εξειδικευμένο θέμα, στο οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία αναφορά. Ε, η έκθεση του συναδέλφου Λάιον είναι πολύ καλή και ιδιαίτερο ισορροπημένη, λαμβάνοντας υπόψη πολλά από τα χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου. Ε, σε ένα θέμα στο οποίο όμως δεν αναφέρεται, είναι η ιδιαιτερότητα που φαίνεται να έχει να αντιμετωπίσει ο νότος Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των κλιματικών αλλαγών, ο οποίος νότος, σύμφωνα με την Επιτροπή, θα πληγεί και πολύ περισσότερο είναι γνωστό ότι οι δραστηριότητες που σήμερα παρουσιάζονται ως εναλλακτικές προτάσεις διαφοροποίησης των γεωργικών δραστηριοτήτων και του γεωργικού εισοδήματος θα συρρυκνωθούν εξαιτία τη αύξηση τη θερμοκρασία, όπω παραδείγματο χάρη δασοκομεία, χειμερινό τουρισμό κτλ. Επομένω, εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση, διότι αφαιρούνται από ορισμένε περιοχέ οι δυνατότητε και να διαφοροποιηθούν εισοδηματικά βελτιώντα τη δυνατότητα προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αλλά και να στραφούν προς την παραγωγή δημόσιων αγαθών, η οποία παραγωγή δημόσιων αγαθών, όπως προτείνεται πολύ σωστά, θα πρέπει να ανταμείβονται. Φαίνεται δηλαδή ότι η κλιματική αλλαγή αποστερεί από ορισμένε περιοχέ τη δυνατότητα να διατηρηθούν ενεργέ οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμες. Αυτό το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί διότι είναι μεγαλύτερος από ποτέ ο κίνδυνος ερημοποίησης αυτών των περιοχών. Και θα πρέπει βέβαια να δούμε με ποιο τρόπο θα επιτευχθεί αυτό χωρίς να δημιουργηθούν νέες στρεβλώσεις, αλλά και χωρίς να, να αποστερήσουμε τη δυνατότητα σε αυτές τις περιοχές να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους. Θα πρέπει να στηριχθούν οι περιοχές αυτές σε συγχρηματοδότηση ή από τον, από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Θα πρέπει να στηριχθούν αυτές οι περιοχές με αποζημίωση για το εγγενές μειονέκτημά τους ή θα πρέπει να στηριχθεί η εισαγωγή άλλων δραστηριοτήτων για διαφοροποίηση. Και βεβαίως ποιε θα μπορούσαν να είναι αυτές οι νέες δραστηριότητες και με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να στηριχθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ανιώ ε, και ρέμες και κλείνουμε. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Ανιώ ή Άγνιο. Μίλησε ο κύριος Επίτροπος για κλιματική αλλαγή πολλές φορές. Αλλά βλέποντας τους δύο τελευταίους ε, χειμώνες που πάγωσε το κοκαλάκι μας δεν είναι αποδεδειγμένη η κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δείχνουν, πολλές ενδείξεις που δείχνουν ότι δεν είναι αποδεδειγμένη η κλιματική αλλαγή. Αλλά ακολουθείς κανείς ένα τέτοιο δρόμο. Τα πράγματα δεν θα είναι θετικά για τους γεωργούς. Αντί να είναι οι καλοί γιατί καταναλώνουν διοξείδιο του άνθρακο στα χορτάρια τους. Φαίνεται τώρα ότι οι αγελάδες τους όταν ρεύονται παράγουν αέρια θερμοκηπίου και είναι τα κακά. Τα κακά παιδιά στην κοινότητα. Και τους κατηγορούμε γιατί χρησιμοποιούν σόγια και όλα αυτά. Λοιπόν, μέχρι ποιο σημείο θα ακούτε αυτούς που λένε όλες αυτές τις ιστορίες και τα παραμύθια για την κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ. Ρέιμερς, ένα λεπτό παρακαλώ. Ακούσαμε λοιπόν ότι η κοινή αγροτική πολιτική θα πρέπει να εκπληρώσει τις προσδοκίες της κοινωνίας. Αυτό είναι όμως μια μεγάλη απέτηση. Και υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος ότι μπορεί να, απο... να απομονωθούν οι γεωργοί, να αποκλίνουν πάρα πολύ από την ε, παλιά δραστηριότητα που είχαν παραδοσιακά. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να εφαρμόσουμε στην πράξη της γεωργικές ε, επιχείρησης δεν θα πρέπει να δώσουμε και στον αγροτικό τομέα το χρόνο και τη δυνατότητα να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους αυτούς που θέλουμε. Και φυσικά θα πρέπει να εξασφαλίσουν και την δυνατότητα επιβίωσής τους. Αυτό σημαίνει το να βλέπουμε το δάσος και όχι τα δέντρα. Σικερέσκη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ δύο σχόλια εάν μου επιτρέπετε. Νομίζω πως είχαμε πολλά επιτεύγματα στο παρελθόν ε, της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής και δεν πρέπει να τα παραβλέψουμε. Βεβαίως υπάρχει ανάγκη μεταρρύθμισης ε, της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, οπότε εντάξει να μιλήσουμε για αλλαγή, αλλά να θυμόμαστε και τα επιτεύγματα του παρελθόντος. Και κάτι ακόμα. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει συνένεση μεταξύ διαφορετικών κρατών μελών και κομμάτων όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Έχουμε μία συνένεση για το πώς θα προσεγγίσουμε τους αγρότες, γιατί οι αγρότες κάνουν πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις, όπως ξέρετε. Eh, λοιπόν, έχουμε μερικά λεπτά τώρα για τον George Lyon, όχι για να απαντήσει σε όλα, αλλά τουλάχιστον ε, μέσα σε δύο-τρία λεπτά να δεις εσύ George να εστιάσεις λίγο τα πράγματα, γιατί έχουμε και μια άλλη έκθεση μετά. Και μετά θα ζητήσω και από τον Επίτροπο να κλείσει. George Lyon, έχει το λόγο. Καταρχήν, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου εδώ σήμερα για τη θετική τους συνεισφορά στη συζήτηση αυτή που κάναμε. Υπάρχουν πολλοί χώροι όπου βλέπω να υπάρχει συμφωνία σε όλη την αίθουσα. Υπάρχουν και άλλοι τομείς όπου χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση και εγώ προσβλέπω σε αυτή τη συζήτηση την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο όπου θα συναντηθώ με τους σκιώδεις εισηγητές για να αρχίσουμε να συζητούμε τα θέματα τα οποία έχουν θίξει εδώ. Ίσως θα πρέπει να διευκρινίσω σε ένα-δύο σημεία γιατί μου τέθηκαν και τέτοια αντίστοιχα ερωτήματα. Αναφέρθηκε το θέμα της λεγόμενης γυμνής γης. Έχουμε ένα πρόβλημα στη Σκοτία και ίσως και στην Νότια Ιρλανδία. Υπάρχουν δηλαδή μεγάλες εκτάσεις που δεν έχουν καμία πληρωμή αγροτική και αυτό φυσικά έχει κάποια μεγάλη επίπτωση στην ικανότητα να μπορούμε να προσελκύσουμε γεωργούς. Αυτό είναι ένα θέμα. Θέσατε ένα άλλο θέμα. Τι γίνεται με αυτούς οι οποίοι είναι ερασιτέχνες γεωργοί, οι οποίοι το κάνουν για την ψυχαγωγία τους, αν θα πρέπει να συμπεριληφθούν για το σύστημα πληρωμών. Επίσης, την κυρία Κανιέτη, την ε, λετωνό συναδελφό μου, ανησυχούσε για την ε, σύσταση να υπάρξει μια σταδιακή εφαρμογή επί τη βάση ιστορικών στοιχείων. Αυτό αφορούσε όμως το σύστημα πληρωμής και όχι τους στόχους του προϋπολογισμού. Δεν θέλω λοιπόν να υπάρξει τροποποίηση ή κατάργηση των ε, κονδυλίων στον προϋπολογισμό που προβλεπόταν να υπάρχει αυτή η μετάβαση για τα παλιά κράτη-μέλη από το παραδοσιακό σύστημα στο σύστημα που βασίζεται στην καλλιεργούμενη επιφάνεια. Νομίζω λοιπόν ότι η συζήτηση μας έχει δώσει πολύ επικοδομητικές ε, ιδέες και προτάσεις και πιστεύω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα προσπαθήσουμε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμφωνία και να έχει ισχυρό λόγο η Επιτροπή μας σε όλα αυτά που θα γίνουν στη Γεωργία μετά το 2013. Ευχαριστώ, Τζόρτζ, που κατάφερες να τα πεις ε, τόσο περιληπτικά. Θυμίζω σε όλους, δίνοντας το λόγο στον Τάσαν Σόλος, θυμίζω λοιπόν ότι η ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών στην έκθεση Λάιον είναι 27 Απριλίου. Η 27 Απριλίου, τελευταία ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών. Ε, έχουμε μεταφέρει νωρίτερα την ημερομηνία γιατί περιμένουμε πολλές, πολλές τροπολογίες. Λοιπόν, ευχαριστώ τον ε, Επίτροπο για την διαθεσιμότητά του και το άνοιγμα πνεύματος που τον διέπει για τη Γεωργία. Δεν θα ρίψω, κινδυνέψω να καταλήξω σε συμπεράσματα σε αυτή τη συζήτηση. Και δεν θέλω να προδικάσω τίποτα γιατί θα γίνει και συζήτηση στην Ολομέλεια. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη δουλειά που έγινε εδώ. Θα βελτιωθεί σίγουρα με τις προτάσεις που θα υποβάλλετε. Αλλά ήδη βλέπετε ποια είναι η διάσταση απόψεων ε, αλλά και οι διαφορές απόψεων για ορισμένα θέματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιο είναι το έργο της Κομισιόν, η δυσκολία του έργου να παντρέψει αυτές τις απόψεις και να παρουσιάσει κάτι το συνεκτικό, κάτι το λογικό λαμβάνοντας υπόψη και όλη αυτή τη διαφορετικότητα των απόψεων. Καταλαβαίνω τις ανάγκες της κυρίας Μαγκίνες που θέλει η Κομισιόν να είναι πιο ακριβής και πιο σαφής και να δίνει και μια κατεύθυνση. Συμφωνώ ότι η Κομισιόν πρέπει να παίξει το ρόλο της. Αλλά αν εμείς ε, καθοδηγήσουμε επακριβώς από την αρχή δεν παραμένει περιθώριο για να ακούσουμε τις απόψεις. Εγώ αποφεύγω να σας δώσω εδώ ακριβή στοιχεία. Όχι γιατί δεν τα σκέφτομαι, τα είχα σκεφτεί ήδη όταν ήρθα εδώ στην ακρόαση. Αλλά πιστεύω ότι το να προτρέχει κανείς με ακριβείς, πολύ ακριβείς απαντήσεις σκοτώνει τη δημιουργικότητα των ανθρώπων που έχουν ιδέες. Γι' αυτό λοιπόν αυτού του είδους οι συζητήσεις είναι πολύ σημαντικές για μένα, όχι γιατί μπερδεύουν παραπάνω τα πράγματα, αλλά γιατί διαπιστε... επικεντρώνουν καλύτερα στους στόχους. Έγιναν ερωτήσεις και σχόλια για τις άμεσες ενισχύσεις. Πώς να αναδιανύμουμε τις άμεσες ενισχύσεις. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί να δώσουμε αυτές τις άμεσες ενισχύσεις και αφού καταλάβουμε γιατί θέλουμε να τις δώσουμε και δεν απαντήσουμε δηλαδή σε αυτή την ερώτηση θα έχουμε πάντα το πρόβλημα του να δικαιολογούμε αυτές τις άμεσες ενισχύσεις στον, στον φορολογούμενο. Εγώ θέλω να, καταλάβουν, ε, να καταλάβει ο κόσμος γιατί ποιους στόχους θέλουμε να προσεγγίσουμε με αυτές τις ενισχύσεις και μετά θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε σε αυτήν την αναδιανομή. Ερωτήσεις που δεν έχουν άμεση σχέση με το μέλλον της ε, ΚΑΠ, αλλά θέλω να απαντήσω. Διμερείς ε, συμφωνίες με τις τρίτες χώρες, και πώς να ελέγξουμε τις εισαγωγές. Η κυρία Χέραντς Γκαρσία το το θέμα. Οι διμερείς συμφωνίες που έχουμε και για τα με τις μεσογειακές χώρες έχουν πάντα τις ε, ρήτρες διασφάλισης για τα φρούτα και τα λαχανικά. Έχουμε πάντα αυτά τα μέτρα που μας επιτρέπουν να προστατευτούμε. Τα κράτη μέλη είναι αυτά που πρέπει να απαντήσουν οι ισπανικές αρχές έχουν τα μέσα για να το κάνουν αλλά πρέπει να τα εφαρμόσουν Τώρα κυρία Γκαρσία Πέρε, σίγουρα όλα αυτά θα ρυθμιστούν με ειδικά νομοθετήματα. Όταν θα έχουμε πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα των εργασιών της ε, ομάδας ε, υψηλού επίπεδου. Το ίδιο και για την ε, τροφιμική αλυσίδα. Αυτά τα λύσουμε πριν από τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ το 2013. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να απαντήσουμε πιο γρήγορα σε ερωτήσεις σαφείς. Τώρα κύριε Ταραμπέλα, θα δούμε τότε τι μηχανισμούς ε, θα έχουμε... Θα δούμε τι μηχανισμούς έχουμε και θα κοιτάξουμε να δράσουμε άμεσα με τους υπάρχοντες ε, μηχανισμούς. χωρίς ε, να υπερβάλλουμε στη χρήση αυτών των μέσων για να μην τα καταστήσουμε και αναξιόπιστα. Εμείς μπορούμε βραχυπρόθεσμα να παρέμβουμε με τους μηχανισμούς που έχουμε στη διάθεσή μας. Για την ερώτηση του κυρίου Ταβαντζή. θα πρέπει όλα να γίνουν σύμφωνα με τις συνθήκες. Πρέπει να διασφαλιστεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη ότι εφαρμόζεται η νομοθεσία και για το θέμα των γεών δεν είναι δικιά μου η υπόθεση, είναι η υπόθεση των, ε, της εσωτερικής αγοράς. Και για τη γη ισχύει αυτή η νομοθεσία. Πρέπει η Κομισιόν να κάνει αυτή την νομική επεξεργασία για να μπορέσουν να ερμηνευτούν σωστά και οι συνθήκες. Το Συμβούλιο έλαβε αποφάσεις αγνοώντας υπάρχουσες νομοθεσίες για την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών μεταξύ των οποίων και τη σχέση. Αυτή είναι η υποχρέωση που έχει η Κομισιόν πάντως από τις συνθήκες. Εντάξει, νομίζω ότι Νομίζω ότι έχω απαντήσει στα ερωτήματα αυτά τα οποία δεν συνάπτονται άμεσα με την έκθεση του κυρίου Λάιον, αλλά με τη συζήτηση που ήθελα να κάνω μαζί σας, θα επανέλθω ενώπιόν σας και σε άλλες ευκαιρίες για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω μου είναι ότι και εσείς θα είσαστε παρόντες στην συνδιάσκεψη που θα οργανώσουμε τον Ιούλιο για να δούμε από κοινού με ποιο τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες ιδέες οι οποίες θα αναδυθούν σε σχέση με την κοινή αγροτική πολιτική. Σας ευχαριστώ και πάλι που με προσκαλέσατε και ελπίζω ότι θα έχω και άλλες ευκαιρίες να έρθω ενώπιόν σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ντάσεν. Διακόπτω για μερικά δευτερόλεπτα για να αποχαιρετήσω τον Επίτροπο γιατί μετά έχουμε το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Σχετικά με τον έλεγχο από τα κράτη-μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή. Πολύ μικρή έκθεση, αλλά πρέπει να γίνει οπωσδήποτε τώρα. Mi Συγγνώμη, συγγνώμη, αλλά... Ε, ε, ε, δεν έχουμε ώρα και μετά έχουμε και τους συντονιστές. Abbiamo l'ultimo Τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη, λοιπόν υπομονή. Κυρίως οι συντονιστές με τους οποίους θα συναντηθούμε ευθύς αμέσως, μάλλον άμα τη λήξη της Επιτροπής. Πρέπει να γνωμοδοτήσουμε σχετικά με την Επιτροπή και την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Και αυτή η πρόταση έχει ως σκοπό να πονήσει έναν κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 291 της Λισαβόνας, να περάσουμε δηλαδή από την επιτροπολογία στους νέους κανόνες της συνθήκης για τις εκτελεστικές πράξεις. Παρακαλώ προσέξτε με, διότι θα το συζητήσουμε τώρα σε ελάχιστα λεπτά, είναι ένα θέμα όμως πολύ πολύ σημαντικό. Σε αυτό το κείμενο που θα σας διαβάσω σε λίγα λεπτά, έχουμε χρόνο μέχρι τις 15 Απριλίου, αν θέλουμε δηλαδή να τροποποιήσουμε ή να διορθώσουμε αυτή την έκθεση. Θα διαβάσω σύντομα. Αγαπητοί συνάδελφοι, με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να αποκτήσει την πλήρη νομοθετική εξουσία στον τομέα της γεωργίας. Πολλές φορές λοιπόν θυμήσαμε ότι είμαστε συνομοθέτες με απόλυτη, σε απόλυτη ισοτιμία με το Συμβούλιο. Η συνθήκη της Λισαβόνας τροποποίησε ρίζικα και τον τρόπο εργασίας της Εκτελεστικής Επιτροπής. Πιο συγκεκριμένα την δια... λεγόμενη διαδικασία επιτροπολογίας η οποία θα πρέπει να αντικατασταθεί από εντεταλμένες πράξεις ή συμπληρωματικές πράξεις και αυτό βάσει των άρθρων 290 και 291 της συνθήκης. Ενώ οι πράξεις κατεχώρηση μπορούν πάντοτε να μπλοκαριστούν είτε από το Συμβούλιο είτε από το Κοινοβούλιο που μπορούν να ανακαλέσουν την εντολή που έχουν δώσει στην Κομισιόν ή να εκφράσουν τη διαφωνία τους, οι, συμπληρω... οι εφαρμοστικές πράξεις δεν επιτρέπουν καμία παρέμβαση. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η Γεωργία καλύπτει τις περισσότερες πράξεις επιτροπολογίας. «1.576 πράξεις επιτροπολογίας πέρυσι πέρασαν από την Κομισιόν. και ορισμένες από αυτές τις πράξεις κατεχώρηση ήταν σημαντικότατες και το Κοινοβούλιο δεν μπορούσε να παρέμβει. Στις σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις τα μέτρα που αφορούν στην ΚΑΠ εγκρίνονται με τις λεγόμενες διαχειριστικές διαδικασίες που δεν επιτρέπουν κανένα, καμία παρέμβαση από το Κοινοβούλιο. Απαιτούν μία ε, σταθμισμένη ε, πλειοψηφία από το Συμβούλιο για να μπορέσει να φέρει αντιρρήσεις στην πρόταση της Κομισιόν. Η πρόταση της Κομισιόν για να ρυθμίσει τις, τα, τις, τις εφαρμοστικές πράξεις της Κομισιόν προβλέπει μία αυτόματη ε, μεταβολή αλλαγή μάλλον των διαχειριστικών πράξεων σε εφαρμοστικές ε, πράξεις. Και αυτό είναι απαράδεκτο για την Επιτροπή μας, διότι θα επιβάρυνε την γεωργική, ε, διάφορους τομείς της γεωργικής πολιτικής, αλλά και θα δημιουργούσε πρόβλημα στο Κοινοβούλιο. Μία αυτόματη προσαρμογή των κατεχώρησιν πράξεων θα μπορούς, μπορεί να οδηγήσει να θεωρηθούν αυτές ως εφαρμοστικές. Πρέπει να γίνει λοιπόν μία διάκριση μεταξύ κατεχώρησιν πράξεων στις οποίες έχει δικαίωμα λόγου το Κοινοβούλιο και εφαρμοστικών πράξεων για τις οποίες δεν έχει κανένα λόγο το Κοινοβούλιο θα πρέπει να γίνεται αναπερίπτωση. Δεν θα πρέπει αυτόματα να μετατρέπονται σε κατεχώρηση πράξης. Προτείνω λοιπόν στη γνωμοδότησή μου να διαγράψουμε το άρθρο 10 της πρότασης της Κομισιόν. Αντί να προτείνουμε μία απαράδεκτη αυτόματη διαδικασία η Κομισιόν θα πρέπει να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατόν τις απαραίτητες νομοθετικές προτάσεις για την προσαρμογή του κεκτημένου χωρίς καθυστέρηση. Το Κοινοβούλιο αντίθετα με το τι θέλει η Κομισιόν θα πρέπει να διατηρήσει τα υπάρχοντα δικαιώματά του διατηρώντας δηλαδή τις ε, πράξεις της επιτροπολογίας εκείνες που πρώτα εντάσσονταν στη διαδικασία συναπόφασης. Μία αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να συμμετέχει στις επιτροπές των εκπροσώπων των κρατών μελών, πράγμα που το κάναμε στην ε, ομάδα υψηλού επίπεδου Γάλα. Συμμετέχει εκεί το Κοινοβούλιο. Υποστηρίζω ότι ως συνομοθέτες το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι σε θέση να φέρουν αντιρρήσεις σε εφαρμοστικά μέτρα τα οποία είναι, αντιβαίνουν στις αρχές της συνθήκης της Λισαβόνας. Και θα πρέπει όλα αυτά να γίνονται μέσα από την εξεταστική διαδικασία. Θα πρέπει να υπάρχει μία διαδικασία εξεταστική διαδικασία η οποία εξεταστική διαδικασία έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τη συμβουλευτική διαδικασία και στην οποία εκτελεστική διαδικασία πρέπει να συμμετέχουν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να αναλάβουμε τη συνομοθετική μας αρμοδιότητα απόλυτα και θα πρέπει να καταστήσουμε αποτελεσματικά και στις νέες εξουσίες που μας χορηγεί η συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν μπορεί η Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίζει για τη Γεωργία χωρίς δημοκρατικό έλεγχο. Και τέλειωσα. Ευχαριστώ. Αυτά. Αυτή είναι η... Αυτό είναι το σχέδιο γνωμοδότησης. Έχουμε τρεις μέρες μέχρι τις 15 του μηνός για τροπολογίες. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ανοίξουμε συζήτηση, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα. Είναι θεμελιώδες να μην προχωρήσουμε στην αυτόματη μετατροπή σε εφαρμοστικές πράξεις. Okay, intanto do la parola ad Albert Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Πάολο, θα είμαι σύντομος. Πλήρης κάλυψη από την ε, ομάδα μας. Δεν μπορεί εδώ πέρα λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς το Κοινοβούλιο. Συμφωνούμε πλήρως ε, με την απόφαση σας εδώ πέρα. Την υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ, Λουίς Καπλασάντος. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, συν συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη του προλαλήσαν. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν θέλει το λόγο. Ένα λεπτό. Γιατί μετά έχουμε και συντονιστέ. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Και μονάχα θα ήθελα να σταθώ στο σημείο του άρθρου 10. Νομίζω ότι υπάρχει μια παρ εξήγηση σε σχέση με αυτό που θέλω να την διαλύσω. Το άρθρο 10 για την αυτόματη ευθυγράμμιση δεν ανατρέπει την ανάγκη ενδεχομένως ορισμένες πράξεις να προσαρμοστούν στο νέο δεδομένο των κατεχώρησης πράξεων. Επομένως, υπάρχουν ορισμένοι χώροι ήδη που στο φως των τωρινών συνθηκών πρέπει να αντιμετωπιστούν από πράξεις κατ' εκχώρηση, αυτό πρέπει να το εξετάσουμε εν ευθέτω χρόνο με τον κατάλληλο τρόπο. Αλλά εδώ δεν αναφερόμαστε στο άρθρο 10. Το άρθρο 10 δεν αναφέρεται αυτό στο άρθρο 10. Το άρθρο 10 προσπαθεί να επιτύχει με ένα αυτόματο τρόπο να μεταφέρει όλες τις επιτροπές στο νέο σύστημα επιτροπολογίας. Άνευ του άρθρου 10 θα παραμέναμε για πολλούς μήνες με μια κατάσταση χαοτική που θα έχουμε μια νέα επιτροπολογία με παλιές επιτροπές συμβουλευτικές, κανονιστικές κτλ. Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα λοιπόν το ότι θα πρέπει να λάβετε υπόψη αυτή την κατάσταση και να μην ζητήσετε την κατάργηση του άρθρου 10. Διαχωρίστε αυτά τα δύο θέματα, αφενός την τεχνική και αυτόματη μεταφορά για να μην υπάρξει χάος και μπάχαλο και από την άλλη μεριά υπάρχει η πολιτική διαδικασία της επαρεξέτασης της ε, υπάρχουσας νομοθεσίας που πράγματι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί για να δούμε ποιες από αυτές τις ε, πράξεις θα πρέπει να είναι μέσα στις πράξεις κατεχώρηση. Ευχαριστούμε την Κομισιόν για την ε, διευκρίνηση. Θα μπορούσε όμως να ξαναγραφεί το άρθρο 10 για να αποφευθούν οι συνθήκες, οι, συγγνώμη, <laughs> οι συγχύσεις και να Αποφευθούν λοιπόν οι παρεξηγήσεις σεβόμενοι τις αρχές της συνθήκη τη Λισαβόνα. Θα ήταν καλό πράγμα λοιπόν, περιμένουμε να ξαναγραφτεί αυτό το άρθρο. Αν δεν υπάρχουν άλλες τοποθετήσει, θα μπορούμε να το ξανασκεφτούμε το θέμα αυτέ τι μέρες γιατί θα το ψηφίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση. Ωραία. λίγοι. Η συνεδρίαση παρακαλώ τους συντονιστές να παραμείνουν για μια συντομότατη συνάντηση χωρίς διερμηνή αλλά θα τα βγάλουμε πέρα. Ευχαριστώ πολύ.